Hello. Hello. Okay. Okay, now it's okay. Good. Um, um, good afternoon. Καλησπέρα σας. Επανερχόμαστε μετά το σύντομο μεσημεριανό διάλειμμα. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Επίτροπο Ελσπιέτα Μπιενκόφσκα, αρμόδια για την ιστορική αγορά, ε, την επιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα συνεχίσουμε το διαρθρωμένο μας διάλογο συμπεριλαμβανομένης και τη συζήτηση ε, για τις ε, πρόσφατα εγκριθήσεις νομοθετικές προτάσεις για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα συζητήσουμε πρώτα απ' όλα, κύριε Επίτροπε, τρία θέματα που είναι σημαντικά. Βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα κινητοποίησεων λόγω της εργασιακής διένεξης με τη διοίκηση για τις συνθήκες εργασίας μας, οι διερμηνείς. Σε ορισμένε καμπίνε έχουν επιστρατευθεί όλοι οι διερμηνεί και είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν. Αυτό καταργεί το δικαίωμα στην απεργία και είναι διάκριση για τι υπόλοιπε γλώσσε. Γι' αυτό, όσο αλληλεγγύη, η ελληνική καμπίνα δεν θα κάνει στάση εργασία που προβλεπόταν. Δυστυχώ όμω, δεν θα παραχωρήσουμε καμία υπέρβαση ωραρίου και θα σταματήσουμε την προβλεπόμενη ώρα λήξης. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε λοιπόν να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιό σα και που είναι και δική μα αρμοδιότητα, όπω επιχειρηματικότητα, μικρομεσαίε επιχειρήσει, ε, ενέργεια, έρευνα. Το θέμα τη άμυνα που σε εμπίπτει στι ε, αρμοδιότητέ μα. Αν και έχουμε κοινή αρμοδιότητα με άλλες επιτροπές στα θέματα άμυνας, αλλά και το πρόγραμμα για το διάστημα που είναι καινούριο και θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για αυτά τα θέματα. Τρία λοιπόν είναι τα βασικά θέματα και είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούμε στην Επιτροπή μας όχι μόνο για την χρηματοδότηση της επόμενης επταετίας, αλλά μας ενδιαφέρει να μας ενημερώσετε πώς βλέπετε τις προοπτικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τη βιομηχανία μας, αλλά και για το πρόγραμμα για το διάστημα και τι μέλλον προβλέπετε στην επόμενη δεκαετία για όλα αυτά τα ζητήματα. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Γνωρίζω ότι σας απασχολεί ιδιαίτερα το επόμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο και παρακολουθείτε διάφορα ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές σας στα πλαίσια του επόμενου ΠΔΠ. Εγώ θα επικεντρωθώ κυρίως στην άμυνα, ε, το διάστημα και το πρόγραμμα της ενία αγοράς, αλλά να πω κάποια εισαγωγικά σχόλια πιο γενικού χαρακτήρα, γιατί όπως ξέρετε κάθε προϋπολογισμός είναι δύσκολος, αλλά ο συγκεκριμένος, ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός ήταν ακόμη πιο δύσκολο ζήτημα. Γνωρίζετε ότι οι δυσκολίε οφείλονται αφενός στο σημαντικό χρηματοδοτικό κενό που θα δημιουργηθεί στο κοινοτικό προπολογισμό λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου έχουμε αύξηση των ε, ε, δαπανών, των αναγκών δαπάνη σε πολλού τομεί, η σε πολλού νέου τομεί, οπως άμυνα. Οπότε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργαζόμαστε εργοδός και επικεντρωνόμαστε στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για να μην ε, ε, φανούμε ανταγωνιστικοί απέναντι σε κάποιες κρατικές δαπάνες. Και γι' αυτό μας απασχολούν ιδιαίτερα οι τρεις άξονες που σας ανέφερα, δηλαδή η άμυνα, το διάστημα και το πρόγραμμα της ενίας αγοράς. Γιατί, γιατί φυσικά στο, στην άμυνα δεν ξεκινούμε εκ του μηδενός. Τα τελευταία χρόνια έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην ε, συνεργασία για την άμυνα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία και το λέω αυτό ως Επίτροπος Βιομηχανίας και για πρώτη φορά στην ιστορία έχουμε ε, αφιερώσει 90 εκατομμύρια ευρώ για μία τριετία ε, για το 2017, 2018 και 2019 9 εκατομμύρια για την ε, έρευνα στην άμυνα και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη. Πέρυσι τον Ιούνιο υποβάλαμε την το πρόγραμμα ανάπτυξης ε, της ε, βιομηχανικής βάσης ε, για τις άμυνες με 500 εκατομμύρια ευρώ για την τελευταία διετία του τρέχοντος ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ για τη διετία 2019 και 2020 και από ό,τι άκουσα σήμερα ψηφίσατε και υπέρ της πολιτικής συμφωνίας στην οποία κατάληξαμε. Οπότε το θέμα θεωρείται λήξαν στο θεωρητικό επίπεδο, θα πρέπει να περάσουμε στην εφαρμογή. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την υποστήριξη που προσφέρει η Επιτροπή σα ε, στα θέματα αυτά και ιδιαίτερε ευχαριστήσει θα ήθελα να απευθύνω στον εισηγητή σα και του σκιώδη εισηγητέ, γιατί πραγματικά μα βοήθησαν ε, ιδιαίτερω στου τριμμένου διαλόγου με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τον επόμενο προπολογισμό. Προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε τι ε, πρωτοβουλίε αυτέ να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα προτείναμε 13 δισεκατομμύρια ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το EDF. Μάλιστα πρόκειται για εξαπλασιασμό του προϋπολογισμού και σε σχέση με τα δύο πειραματικά προγράμματα στο τρέχον ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτό που έχουμε προσφάτως συμφωνήσει. Επαναλαμβάνω, δεν ξεκινούμε εκ των μηδενός, γιατί και πειρα έχουμε και αποτελέσματα έχουμε. Οπότε μαζί με, την, με το νέο τομέα ασφάλειας και άμυνας, γιατί προτείνουμε νέο τομέα ε, στον επόμενο προϋπολογισμό που θα αφορά την ασφάλεια και την άμυνα και εκεί έχουμε 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στρατιωτική κινητικότητα και ελπίζω ότι προβλέπουμε επαρκή χρηματοδότηση για να υλοποιήσουμε τους πολιτικούς στόχους της άμυνας. Και μάλιστα έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει ο τέταρτο επενδυτή σε θέματα άμυνα ε, στην Ευρώπη και φυσικά το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο θα είναι το βασικό όργανο στήριξη τη αμυντική συνεργασία στην Ευρώπη. Και εμεί ε, θα στηρίξουμε όλη την, όλη την, την αλυσίδα αυτού του κλάδου, από το σχεδιασμό μέχρι την δημιουργία ικανοτήτων. Δεύτερη φάση είναι η έρευνα. 4,1 δις προβλέπεται γι' αυτό, έρευνα στην άμυνα και είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι σε αυτό το τμήμα του προγράμματος τα διάφορα σχέδια θα λάβουν πλήρη και άμεση χρηματοδότηση, πλήρη επαναλαμβάνω και άμεση χρηματοδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Στόχος μας εδώ είναι πραγματικά να γεφυρώσουμε το τεχνολογικό χάσμα και να βοηθήσουμε την Ευρώπη να καλύψει αυτό το τεχνολογικό κενό. Δεύτερο στάδιο, ανάπτυξη ε, αμυντικών ικανοτήτων, 8,9 δις. Εδώ θα συγχρηματοδοτήσουμε 20% του συνολικού ε, κόστους της ανάπτυξης πρωτοτύπων και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν το 80%. 20% θα πάει από το κοινοτικό προπολογισμό και 80% από του εθνικού προπολογισμού. Άλλο βασικό στοιχείο των ταμείων είναι 5% του προπολογισμού θα αφιερωθεί στην ε, στήριξη των ε, disruptive technologies ε, και σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική βάση για την άμυνα, απαιτούμε τουλάχιστον τρει εταιρείε από τουλάχιστον τρία κράτη-μέλη και θα συγχρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη πρωτοτύπων μόνο όταν τα κράτη-μέλη δεσμεύονται να αγοράσουν από κοινού τα τελικά προϊόντα. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε επιδοτήσεις, αλλά θα προβλέψουμε και τη δυνατότητα για προεμπορική ε, κρατική προμήθεια, όπως γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Και θέλουμε, όπως γίνεται και με την βιομηχανική βάση για την άμυνα, να εθαρρύνουμε την ε, συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ε, επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, mid-caps, γιατί είναι πολλές οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Και το διασυνοριακό σκέλος είναι πολύ σημαντικό, οπότε θα δώσουμε ένα ειδικό μπόνους και ένα επιπλέον κριτήριο για αυτούς. Ο στόχος είναι σαφής. Θέλουμε να ανοίξουμε την Ευρωπαϊκή Αλυσίδα Αξίας. Γιατί τα κονδύλια δεν είναι μόνο για τις μεγάλες χώρες μέλη και τις μεγάλες επιχειρήσεις, είναι για όλους για όλα τα κράτη-μέλη και για τις μικρομεσαίες και για τις μεσαίες κεφαλαιοποίησεις επιχειρήσεις. Επίσης, έχουμε κάποια συνέργεια με τα σχέδια της ΠΕΣΚΟ και αυξανόμενη χρηματοδότηση για μεγαλύτερη ικανότητα των σχεδίων της ε, ε, ΠΕΣΚΟ. Τώρα, ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι το κριτήριο επιλεξιμότητας, δηλαδή ποιο μπορεί να έχει πρόσβαση ε, σίγουρα η συμφωνία που έχουμε με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την EDIP, την ε, βιομηχανική βάση για την άμυνα, θεωρώ ότι θα, θα λάβει χώρα γιατί η πρόταση είναι ισορροπημένη και διευρύνει τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ, αποφεύγοντας επικαλύψεις και διαφυλάσσοντας ε, τα συμφέροντα ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπολογίζω στη δική σας υποστήριξη για να ε, προωθήσουμε τις φιλοδοξίες μας και είμαι ήδη έτοιμη να ξεκινήσουμε τις εργασίες με τη νέα διαπραγματευτική σας ομάδα. Είμαι στη διάθεσή σας. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σημείο, ε, πολύ σημαντικό θέμα, το διάστημα. Πριν από δύο εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 16 δις για το πρόγραμμα, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το Διάστημα όπως ξέρετε πριν από πολλούς μήνες, από 1,5 χρόνο, είχαμε υποβάλει τη στρατηγική του διαστήματος και τώρα με την πρόταση του προγράμματος δίνουμε το όραμα και τις φιλοδοξίες, δίνοντας άρκα και οστά στη στρατηγική μας με συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να κρατήσουμε την πρωτοκαθεδρία μας παγκοσμίως στο διάστημα. 16 δις, ε, καθόλου αμεληταίο ποσό και δώσαμε μάχη για να ε, προταθεί ε, δεν, συμπεριλαμβα... δεν συμπεριλάβαμε ακόμη τα χρήματα από την έρευνα του διαστήματος, αλλά ήδη ε, προτείνουμε σημαντική αύξηση σχέση με τον τρέχοντα προϋπολογισμό για το διάστημα και αυτό είναι μείζον επίτευγμα κατά τη γνώμη μου. Οπότε έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι από τα μέχρι τώρα επιτεύγματά μας στα προγράμματα διαστήματος και είναι το επίτευγμα κοινοτικό, κοινό, όχι ενό κράτου μέλου μόνο. Έχουμε το Κοπέρνικο, το Γαλιλαίο, που είναι πραγματικά πρώτη τάξη υποδομέ και συστήματα. Και επίση ε, είναι πολύ έγκαιρη η εφαρμογή τους και τηρήθηκαν και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί για αυτά. Για την επόμενη επταετία η πρότασή μου είναι σαφής. Συνέχεια εξέλιξη και προσαρμογή. Συνέχεια. Πρωταρχικός στόχο είναι να διατηρήσουμε και να αναβαθμίσουμε υπάρχουσες υποδομέ. το Γαλιλαίο, το Έγνο και το Κοπέρνικος, γιατί η συνέχεια στο διάστημα, στην πολιτική διαστήματος είναι το παν θα πρέπει να διατηρήσουμε ό,τι χρειάζεται να μείνει και να το αναβαθμίσουμε ό,τι χρειάζεται βελτίωση. Για το Γαλλίο και το Έγνος προτείνουμε 9 συν 7 δις επενδύσεις για να συμπληρώσουμε την υποδομή και να προετοιμάσουμε τη δεύτερη γενιά του συστήματος με στόχο να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη στη διαχείριση κυκλοφορίας, σε αυτόνομα αυτοκίνητα, προκειμένου να αναπτύξουμε την στρατηγική μας για την ασφάλεια ταυτόχρονα. Για το Κοπέρνικος έχουμε 5,8 δις, γιατί είναι το πιο προηγμένο σύστημα παρακολούθησης ε, ε, στον κόσμο και θέλουμε να διατηρήσουμε την αυτονομία μας ε, και το μελλοντικό καθήκον για το Κοπέρνικος θα είναι η ευρωπαϊκή ασφάλεια και η ευρωπαϊκή ηγετική θέση για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Επίσης θα κρατήσουμε δύο αποστολές ε, στην πολική ζώνη και θα προσθέσουμε μια εφαρμογή ασφάλειας στον Κοπέρνικο. Τα δεδομένα του Κοπέρνικος θα είναι ανοιχτής και ελεύθερης πρόσβασης δωρεάν και ελεύθερης πρόσβασης. Όλε οι εταιρείε μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τους προσφέρουμε δωρεάν και ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα του Κοπέρνικους. Δεύτερη προτεραιότητα είναι η προσαρμογή στις νέες, στη νέα πραγματικότητα. Και από αυτή την άποψη το διάστημα θα πρέπει να προωθηθεί γιατί είναι προϋπόθεση για την ασφάλεια, θα διευκολύνει την ασφάλεια και γι' αυτό έχουμε δύο νέες πρωτοβουλίες με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ. Η κατάσταση ε, επαγρύπνησης για το διάστημα και Gov.com, κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες. Φυσικά για το διάστημα δεν υπάρχει ε, ευρωπαϊκή αυτόνομη πολιτική με αυτόνομη ε, πρόσβαση, αλλά θέλουμε μια μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα, προβολή και βιωσιμότητα στους εκτοξευτήρες μας, όπως είναι η Αριάν 6 και ο Vega C. Και επίση θέλουμε να στηρίξουμε τα χρήματα αυτά την ανάπτυξη της ε, χερσαία υποδομή. Και με το ορίζοντα Ευρώπη θέλουμε να έχουμε ένα είδο GTI διαστημική εταιρική σχέση που θα επικεντρωθεί κυρίω στι ρηξικέλευτες τεχνολογίες, τι Raptive Technologies. Επίση προωθούμε τη νέα διαστημική προσέγγιση για την Ευρώπη για καινοτόμε και ρηξικέλευτες νεοφυεί επιχειρήσει που ενεργοποιούνται στο διάστημα. Πέραν αυτού του διαστημικού προγράμματος έχουμε να προτείνουμε κάποια προσαρμογή της διακυβέρνηση με την υπηρεσία διαστήματος επιτροπής και τις υπηρεσίες μας της Πράγας στην GSA και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα αυτό θα ονομαστεί η νέα υπηρεσία για το διαστημικό πρόγραμμα και το μήνυμα που θέλω να σας δώσω είναι ότι δεν αλλάζουμε την ισορροπία των αρμοδιοτήτων δεν αφαιρούμε αρμοδιότητες από κάποια υπηρεσία, θεσμικό όργανο. Η υπηρεσία διαστήματος θα, συνεχίσει να είναι ο κυρίως αρμόδιο το εθνικό πρόγραμμα και η υπηρεσία της Πράγας θα συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει και σήμερα. Αλλά βέβαια σας τονίζουμε ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί ιδίω όσον αφορά την ασφάλεια. Αυτό που θα παρουσιάσουμε στοχεύει στην εξέλιξη και όχι σε κάποια επανάσταση και ελπίζουμε ότι μπορεί να πολύ θετική σα βοήθεια για τα διαστημικά προγράμματα. Πρόκειται για κάποια φιλοδοξία ε, που αφορά τον προπολογισμό, τις δραστηριότητες και είναι πολύ σημαντική πολιτική για την οικονομία μας. Επίσης, μακρηγόρησα, αλλά είχαμε αυτά τα τρία σημεία, τα τρία προγράμματα και όσον αφορά την ενιαία αγορά και το σχετικό πρόγραμμα, ένα από τα μαθήματα. Ήταν 25η επέτειό τη. και όλα αντλήσαμε το συμπέρασμα ότι η ενιαία αγορά είναι κάτι παραπάνω από έναν κανονισμό ε, χρειάζεται υλοποίηση, χρειάζεται εφαρμογή και όλα αυτά τα χρόνια είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιο είδους εργαλεία πιο ήπια, ε, ξεκάθαρη ενημέρωση, πρακτική παροχή συμβουλών, χρηματοδότησης της ΜΜΕ και να από δύο εβδομάδες κατεβάσαμε ένα καινούριο πρόγραμμα σε καινούριο πλαίσιο για πολλές δραστηριότητε και αυτό χωρίς γραφειοκρατία λοιπόν πιο, ε, πιο αποτελεσματικό διότι τέσσερα δίστανε τα για τις ε, νεοφυείς, για τις ΜΜΕ επί τη βάση ε, των επιτυχιών του κόσμου οπότε έχουμε και το Enterprise Europe network, ένα δίκτυο το οποίο αφορά κάποιες υπηρεσίες που παρέχονται ούτως ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ε, τους κανόνες της ενιαίας αγοράς. Να υπάρχει κάποια εποπτεία και για τα οχήματα με κινητήρα, προστασία του καταναλωτή, ασφάλεια για τα προϊόντα και να συνεχίσουμε την παραδοχή ενημέρωσης και συμβουλών για την ενιαία αγορά και επίσης για αυτό που σημαίνει για τον τελευταίο μήνα όσον αφορά τα ψηφιακά, την ψηφική λεωφόρο και να έχουμε επίσης προτυποποίηση και προστασία των καταναλωτών. Όλες αυτές οι δραστηριότητε θα ενταχθούν ε, σε αυτό το πλαίσιο του προγράμματος των 4 δις για την ενιαία αγορά. Και σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου διαθέσατε ο Πρόεδρος. Πολύ σας ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Να αρχίσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Κρασνοντέμψκι είναι ο εισηγητής μας για το πρόγραμμα άμυνας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Επίτροπε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που καταφέραμε να συνεργαστούμε στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα σε κάποια θετικά σημεία του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φαίνεται από αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη πάρα πολλές προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έλαβε υπόψη και το αποτέλεσμα των τριμερών διαπραγματεύσεων σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική βάση για την άμυνα, η DIDP. Απαιτείται δηλαδή ε, απαιτούνται τουλάχιστον τρεις εταιρείε από τουλάχιστον τρεις ε, χώρες μέλη. Συμμετοχή ε, μικρομεσαίων και μεσαίων κεφαλαιοποίηση επιχειρήσεων. Δυνατότητα χρηματοδότηση και μη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εφόσον έχουν έδρα και σε ευρωπαϊκές χώρες. Και επίσης ε, δίνονται κίνητρα για χρηματοδότηση διασυνοριακής συνεργασίας, ε, κάποια τεχνολογικά ζητήματα που θα ε, συμπεριληφθούν στη συζήτηση αργότερα. Και μετά τα θετικά να αναφερθώ και σε κάποια αρνητικά σημεία. Κατά τη γνώμη μου, το πιο αρνητικό σημείο είναι γιατί δεν περιμένατε ε, να συγκεντρώσετε εμπειρίες από την EDIDP. Αυτή η βιασύνη, αυτή η σπουδή, κατά τη γνώμη μου, το μείζον αρνητικό σημείο. Η ιδέα της ε, EDIDP είναι να δοκιμάσει κάποιες λύσεις. Ενώ το να βελτιώσουμε την ε, λειτουργία του Ταμείου, ενώ μόλις έχει αρχίσει να λειτουργεί, είναι υπερβολικά εσπευσμένο κατά τη γνώμη μου και βεβαιασμένο. Κρίμα που δεν ε, διευκρινίστηκε περισσότερο αυτή η διαδικασία. Ένα άλλο θέμα είναι αυτό το 60% που προτείνει ως ποσοστό χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. δεν είναι αρκετό αυτό το ποσοστό γιατί πρόκειται για μεγαλεπίβολα σχέδια. Οπότε ένα τόσο χαμηλό επίπεδο σε χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ίσως αποθαρρύνει ε, κάποιες επιχειρήσεις να λάβουν μέρος. Κάτι άλλο που αναφερθήκατε, στο οποίο αναφερθήκατε κι εσείς, αλλά σίγουρα θα συζητηθεί περαιτέρω, είναι το θέμα της διαχείρισης των σχεδίων με τη συμμετοχή κρατών μελών στη διαδικασία. Γιατί η αρχή της διπλής επιτροπολογίας ε, ε, υιοθετήθηκε ε, μόνο για ε, προγράμματα, για την επιλεξιμότητα προγραμμάτων που αναφέρονται σε ικανότητα και όχι μόνο σε ερευνητικά προγράμματα. Οπότε, πρώτη, πρώτη ερώτηση, προς τι αυτή η βιασύνη. Γιατί δεν περιμένουμε λίγο να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και μετά από τα συμπεράσματα που θα αντιλήσουμε και από τις εμπειρίες αυτού του δοκιμαστικού προγράμματος του EDIDP, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Και για το ε, Ταμείο Άμυνας, μάλλον, ναι, ως προς το, ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Επίσης, ε, τι γίνεται με την Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου, γιατί υπήρχαν, υπήρξαν κάποια προβλήματα. Και το πρόγραμμα EDL, πώς θα συνδυαστεί με άλλα προγράμματα, με τον Ορίζοντα Ευρώπη, για παράδειγμα. Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια, και για αυτό το θέμα. Πώς θα λάβει χώρα αυτή η συνεργασία, πώς θα συνδυαστούν ή πώς θα εξασφαλιστούν συνέργειες μεταξύ των επιμέρους προγραμμάτων. Αυτά ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κρασνοντέμσκι. Ο κύριος Κρασνοντέμψη, όπως είπα, είναι ο εισηγητής για το θέμα αυτό της Επιτροπής ΣΥΤΡΕ. Και τώρα περνάμε στους κοιόδης ηγητές εκ μέρους του ΕΛΚ. Το λόγο έχει η κυρία Γκροστέτ. Ε, εδώ είμαι κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε δεν άκουσα αμέσω το όνομά μου. Κυρία Επίτροπε, πρώτα σας ευχαριστώ που ήλθατε να μας δείτε. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να συζητούμε μαζί σας για τόσο σημαντικά άλλωστε θέματα. Θα ήθελα με την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω επίσης για την βοήθεια που προσφέρατε εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλες τις εργασίες που έχουμε διεξαγάγει ως τώρα σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα ώστε να προλάβουμε να φτάσουμε σε συμφωνία στους τριμερείς διαλόγους για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αμήνης μεγάλη και πολύτιμη βοήθεια σας. Τώρα για την άμυνα. 13 δισεκατομμύρια για να ενισχυθεί η κοινοτική προσέγγιση για τους εξοπλισμούς. Αυτά ανταποκρίνονται στις ανησυχίες των πολιτών, αλλά και στην ανάγκη αποδοτικής χρήσης του προϋπολισμού και βελτιωμένης συνεργασίας μεταξύ των χωρών μελών. Για τα θέματα αυτά είναι γνωστό ότι υπάρχει και μια, ένα, μια αντίδραση των χωρών μελών που τίνουν προς την ε, διακυβερνητική συνεργασία. Τι μπορείτε να κάνετε για να εξασφαλίσετε μια κοινοτική προσέγγιση για την διαχείριση του εν λόγω ταμείου. Διαχείριση που είναι ένα πραγματικό θέμα. Και πώς ε, να προτρέψετε τις χώρες μέλη που ε, ε, να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα όσα θα ενισχύσει το ε, Ταμείο. Τώρα για το διάστημα. Βέβαιως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει πραγματική διαστημική δύναμη. Έχω κάποιες αμφιβολίες τώρα σε ό,τι αφορά πρώτα την υποστήριξη για το πρόγραμμα Gotras.com για την ασφαλή πρόσβαση που μου φαίνεται ωστόσο με 250 εκατομμύρια σε 7 χρόνια μου φαίνεται κάπως υποχρηματοδοτούμενο. Είναι κάπως απογοητευτικό αυτό. Είναι σοβαρό να, επιμένει κανείς σε αγορά αμερικανικής τεχνολογίας. Δεν δείχνει κάποια έλλειψη για το δικό μας πρόγραμμα θεωρώ ότι θα έπρεπε να διευρυνθεί ο προπολογισμό αυτό και το ίδιο για την πρόσβαση στο διάστημα. Και τελειώνω, είναι θεμελιώδε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να συγκεντρώσει την ε, θεσμική προσέγγιση, τη ε, θεσμική ζήτηση, ώστε να ενισχύσει την κοινοτική διάσταση σε ό,τι αφορά και την απασχόληση αλλά και την αυτονομία, δίνοντας μια ξεκάθαρη υποστήριξη στο, στην συγκέντρωση των προσπαθειών για, τους, ε, για τα οχήματα που θα μεταφέρουν τους δορυφόρους στο διάστημα. Σε ευχαριστώ. Ακολουθεί ο Σκιώδης συγητής για τα προγράμματα μήνης. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς κυρία Επίτροπε που προσήλθατε ενώπιον της Επιτροπής Βιομηχανίας για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμήνης. Δεν θα επανέλθω στη συζήτηση που διεξήθηκε για τον τριμερή διάλογο. Δεν χρειάζεται γιατί τα είπαμε αυτά. Παράταση λοιπόν της πρώτης αυτής δράσης. Εδώ έχω τρεις ερωτήσεις για τη νέα πρόταση. Πρώτα, εκτελεστικός οργανισμός για τη διαχείριση του Ταμείου. Θα αλλάξει τον ρόλο του διακυβερνητικού οργανισμού αμήνης και πώς θα διαρθρώνονται οι ε, δράσεις τους. Δεύτερη ερώτηση. πραγματικά ελέγχθηκε από τον διπλανό μου προηγουμένως και δικαιολογείται από το επίγον του προβλήματος ότι υπάρχει μια διαδοχή ανάμεσα στα προηγούμενα μέτρα που μόλις ψηφίσαμε και στην ίδρυση ενός νέου ταμείου. Και έχουμε πράγματι ένα πρόβλημα αξιολόγησης. Να αξιολογηθούν δηλαδή τα αποτελέσματα του πρώτου σχεδίου. Υπό τις συνθήκες αυτές θεωρείται ότι μια ενδιάμεση αναθεώρηση της επόμενης φάσης θα είναι δυνατόν, θα είναι εφικτή για να διορθωθούν ενδεχομένω κάποιες ελλείψεις. Τέλος, πώς βλέπετε τον σύνδεσμο μεταξύ των 6,5 δισεκατομμυρίων της στρατιωτικής κινητικότητας που εντάσσονται στην διασύνδεση για, την, για διευκόλυνση για τη διασύνδεση Ευρώπης και εάν υπάρχει μια θεματική ενότητα γιατί βέβαια τα 6,5 δισεκατομμύρια είναι σημαντικός προϋπολογισμός. Τέλος, για το διάστημα. Σας συγχαίρω για την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα επανέλθω στα δορυφορικά δίκτυα. Φάνηκε πόσο δεν είναι ικανές οι χώρες μέλη να αναλάβουν την ελάχιστη δυνατή δράση στα θέματα αυτά. Για την πολιτική των εκτοξευτήρων επανέρχομαι στην ερώτηση κυρίας Γκροστέτ. Η πρόσβαση στο διάστημα είναι ζήτημα κυριαρχίας, απόλυτα θεμελιώδες και εξελίσσεται σημαντικά. Και με την παρεμβολή του ιδιωτικού τομέα για και όχι μόνο για την Κίνα και για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Θα θεωρηθεί λοιπόν η κοινοτική παρέμβαση ως ε, αναπόσπαστο μέρος της ε, προσέγγισης της, της Ένωσης. Thank you very much, colleague. I... Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Συνάδελφε Μαρδέ, και εσείς είστε για το αμυντικό πρόγραμμα σκιώδης ηγητές. Έχετε το λόγο. Κύριε Μπουζέρ γιατί να μα ε, ζητείτε συγγνώμη, δεν πειράζει, δεν έχω πρόβλημα εγωιστικό. Απλώ φοβόμουν να μην με ξεχάσετε. Γιατί δεν να πω, είμαι σχεδόν συγκητή από την Ιωνία, να εδώ είμαι. Στο φω. Τέλο πάντων, για αυτό με το οποίο ασχολούμαι θα θέλω να πω ότι επαναλαμβάνω την υποστήριξή μου στις κινήσεις των διερμηνέων, γιατί υπάρχουν κάποιες μέθοδοι αντιδημοκρατικές. Έχουν επιστατευτεί οι διερμηνείς και εκδηλώνουν την ε, ελεγγύη μητρό αφορά το Ταμείο Άμυνας. Τα είπε η κυρία Γκροστέτ παρόλα αυτά όμως, το ότι είναι νέο ταμείο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια διαφορετική πολιτική. Και ευχαριστώ κύριε Μιγκόφσκι, ήθελα να δω ποια ε, που είναι τα κριτήρια της επιλεξιμότητας. Τι γίνεται όταν υπάρχει εταιρική σχέση με τρίτη χώρα ή τι γίνεται για τις χώρες Ευρώπης. Θα πρέπει να έχουμε κάποιο είδους εξασφαλίσεις, θα πρέπει να έχουμε ένα καθεστώς στεγανό για τις θηγατρικές των μεγάλων εταιριών. Να μην ως πάρουν άλλοι τις ιδέες και την πρωτοπορία. Επίσης, τι γίνεται με τις εξαγωγές δεν υπάρχει πολιτική κατασκευή όπλων όταν δεν υπάρχει προσανατολισμό εξαγωγικό. Οπότε ίσω και αυτό το μήνυμα αφορά οι και συνεισηγητέ και όλοι οι να δούμε πώς θα μπορούμε να έχουμε κατάλογο χωρών με τι οποίε μπορούμε να κάνουμε τέτοιο εμπόριο και αυτές που δεν πρέπει να κάνουμε. Από τις να είμαστε προσεκτικοί. Μίλησε και εσείς για διοντολογία. Προσοχή στα ρομπότ πολεμιστές. Να μην συσχετιστούν με το ταμείο αυτό. Επίσης, η διακυβέρνηση όσον αφορά αυτό το ταμείο. Θα πρέπει να καταλήξει να είναι αμυντική πολιτική. Άρα να δούμε πώς θα εξοπλίσουμε με αυτή την πολιτική τις ευρωπαϊκές χώρες. Θα πρέπει να πιάσουν τόπο αυτά τα 13 δις. Καινοτομία, παραγωγή, εδώ στην εσωτερική αγορά πρώτα πρώτα. Να η αιρεσιμότητα και η επιλεξιμότητα. Η παροχή 27 ευρωπαϊκές χώρες. Η ιστορική αγορά, είναι ενδιαφέροντα αυτό το οποίο είπατε και θέλω να πω κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι στο χαρτοφυλακείο σας. Θεωρώ και το λέω και το ξαναλέω ότι η εσωτερική αγορά μας έχει στριμώξει μέσω των ίδιων μας των διατάξουν, γιατί είχε απαγορεύσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να γίνουν γίγαντες στο εμπόριο, στον ε, διεθνή ανταγωνισμό. Λόγω των περισσότερων που υπάρχουν και έτσι γίνονται πολύ ευάλωτες. Είναι στρατηγικός ο τομέας. Και θα πρέπει οι κανόνες μας να επιτρέπουν στην ευρωπαϊκή βιομηχανία να θωρακίζεται σε σχέση ας πούμε με τους κινέζικους ε, σιδαδρόμους και τους άλλους ε, Αμερικανούς γίγαντες. Ε, ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Και παρακαλώ, επόμενο σκιώδες. Για το αμυντικό πρόγραμμα είναι η κυρία Σεβαλία για το ΙΝΕΦ. Και όταν περάσουμε στα υπόλοιπα προγράμματα για το αμυντικό πρόγραμμα, κυρία. Ευχαριστώ. Κυρία Επιτροπέ, εστεριζόμαστε την επιθυμία σας να ενισχύσουμε τη διαλειτουργικότητα των στρατών των ευρωπαϊκών χωρών και να ε, περιορίσουμε την εξάρτησή μας στρατιωτική από τις ΗΠΑ. Πολιτείες. Αλλά αυτό, όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν στα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ ελεύθερων εθνών, όχι με στόχο να καταλήξουμε σε έναν ευρωπαϊκό στρατό. Επίσης, ε, ε, πίσω από τη βούλησή σας για συνεργασία κρύβεται η επιθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταστήσει αλληλεξαρτημένους αυτούς τους κλάδους των κρατών μελών. Και μάλιστα ο πρόεδρος Γιουνκέρ μίλησε για την κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Άμυνας ως βασική πρόπτυγη, κάτι που επιβεβαιώνει τους κρυφούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της Ένωσης ε, Κυρίαρχων και Ελεύθερων Εθνών, μια κυρίαρχη πολιτική υπέρ της Ευρωπαϊκής Άμυνας θα ήταν ένα μέσο που επιτρέπει την τεχνολογική πρόοδο και ε, την ελεύθερη επιλογή της στρατιωτικής συνεργασίας. Η πρόταση σας όμως ε, διευρύνει ε, τις ε, αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον κοινοτικό προϋπολογισμό, περιορίζοντας και συρρυκνώνοντας τις εθνικές αρμοδιότητες. Οπότε δεν θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, γιατί τελικά η χρηματοδότηση θα μπορέσει να ε, ευνοήσει και έξω κοινοτικές επιχειρήσεις, αρκεί να έχουν θηγατρική ε, στην Ευρώπη και να υποφεληθούν από τα αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα για το διάστημα, μας παρουσιάσετε τη φιλοδοξία σας και χαίρομαι που έχετε αντιληφθεί τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι δεν προτείνεται κάποιες στοιχειώδεις λύσεις για να εξασφαλιθεί ε, η διαχρονικότητα αυτού του στρατηγικού τομέα. Γιατί αντιμετωπίζουμε όλο και πιο λυσαλαίο και μερικές φορές αθέμητο τον ανταγωνισμό στο τομέα αυτό. Και εσείς προτείνετε μία, έναν ιωστό οργανισμό που θα καταστήσει ακόμη πιο περίπλοκη την διαδικασία λήψη αποφάσεων, αλλά και θα πετύσει αύξηση του προπολογισμού. Αυτό που θέλουν οι βιομηχανοί, ε, όπω και ο Γενικό Διευθυντή του Αριάν, θέλουν περισσότερη προστασία και αλληλεγγύη από τα κράτη-μέλη. Είναι προφανής οι δύο προτάσεις. Καταρχήν, ε, υποχρέωση χρήσης των ευρωπαϊκών εκτοξευτήρων και την υποχρέωση της, ε, των υπηρεσιών του Γαλλιλαίου για όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα που πολλούνται και χρησιμοποιούνται ε, στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια όταν χρησιμοποιούν τον, την, τον εντοπισμό, τον γεωγραφικό εντοπισμό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λουσία Βαλιέ. Ας μεταφέρετε ομαλά στο δεύτερο πρόγραμμα για το διάστημα. Ας περάσουμε τώρα στο πρόγραμμα για το διάστημα. Περνάμε στον πρώτο νοσομιλητή που είναι ο σκιώδης ε, το ECR για το πρόγραμμα για το διάστημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επίτροπο Μπιενκόφσκα για την παρουσίαση που μας έκανε για το δημοσιονομικό πλαίσιο και τις προτάσεις για τη χρηματοδότηση του προγράμματος για το διάστημα. Το πρόγραμμα διαστήματος είναι ένα από τα μείζωνα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλύπτει μάλιστα όλα τα κράτη-μέλη. Ε, κάτι τέτοιο δεν, να, δεν μπορεί να κάνει κανένα κράτος ε, μόνο του. Θα πρέπει όλα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα για το διάστημα. Ε, με ικανοποιεί και ο προπολογισμό, γιατί σε σχέση με το Γαλλέο και το Κοπέρνικος έχουμε αύξηση των κονδυλίων. Κάτι που δείχνει τη σημασία που έχει το πρόγραμμα για το διάστημα μια ναι, και μπορεί να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπάθησα να βρω μια πιο ε, διεξοδική περιγραφή για τα θέματα αυτά, αλλά δεν τα κατάφερα. Δεδομένης της ε, ε, μεγάλης σημασίας που αρχίζει και αποκτά ο οργανισμός και μάλιστα δεδομένης πρόθεσης να τον μετονομάσετε κάτι που με βρίσκει σύμφωνο, γιατί ο οργανισμός αυτός, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, υποχρηματοδοτείται. Και έχουμε όλο και περισσότερες απαιτήσει από αυτό και αυξάνονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του οργανισμού, αλλά θα χρειαστεί και αύξηση του, των ανθρωπίνων πόρων του ανθρώπινου δυναμικού. Σκοπεύετε να αυξήσετε τον προϋπολογισμό και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Η δεμή θα δημιουργήσει πρόβλημα στην περαιτέρω ανάπτυξη. Μάλιστα. Και περνάμε στο τρίτο θέμα που ανέφερε η Επιτροπός στην ομιλία της, το νέο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά και κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σκιώδης ηγητής της Επιτροπής μας για το θέμα αυτό εκ μέρους του ΕΛΚ είναι ο κύριος Πολ Ρουμπίχ. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για μας όλες και όλους είναι σημαντικό που βλέπουμε ότι η ισχύ της Ευρώπης εξαρτάται κυρίως από το πώς θα πηγαίνουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και βεβαίως αυτές πρέπει να υποστηριχτούν. Όλοι γνωρίζουμε ότι το scaling up και η αλυσίδες δημιουργίας αξίας είναι τα πραγματικά θεμέλια για την θετική εξέλιξη των φορολογικών εσόδων εν τέλει και επομένως και την ικανότητα της Ευρώπης να διατηρεί τα κοινωνικά συστήματα που, στα οποία έχει την πρωτοπορία παγκοσμίω και θα πρέπει να υποστηριχτούν. Γι' αυτό το πρόγραμμα COSME για μένα αποτελεί σημαντική πρόκληση να καταδειχτεί δηλαδή ότι όντως διακατεχόμεθα από την βούληση να ενισχύσουμε νέες ιδέες, καινοτόμες ιδέες για να μπορέσουν να δραστηριοποιούνται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και απασχόληση στην Ευρώπη και ιδίως σε χώρες όπου η ενέργεια των νέων, <clears throat> η είναι υψηλότατη. Το πρόγραμμα COSME μπορεί να παίξει πρωτοπόρο ρόλο εν προκειμένου. Για το Ταμείο Αμήνης και Διαστήματος, ειδικά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση λόγω του ότι προωθούν καινοτόμε λύσεις. Και κόσμε και έγνους και άλλα προγράμματα μπορούν να εφαρμοστούν, τα οποία μας δίνουν την ευκαιρία για το μέλλον να ξαναγίνουμε το νούμερο ένα η Ευρώπη έχει ιστορία αιώνων ως νούμερο ένα. Η γεωπολιτική κατάσταση γύρω από την Ευρώπη, αν την εξετάσει κανείς, αντιλαμβάνεται ότι είναι απολύτως αναγκαίο να ενισχύσουμε τις ικανότητές μας σε αυτόν τον τομέα. Και πιστεύω ότι δύο στις νέες χώρες μέλη υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες, διότι εκεί η τεχνολογική εκπαίδευση ήταν πάντοτε εξαιρετική. Εδώ ανοίγονται νέες δυνατότητες. Ακούσαμε το πρωί ότι ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει να τοποθετεί στρατιωτικές δυνάμεις στο διάστημα. Βλέπουμε ότι αναπτύσσουν τρόπους καταπολέμησης ή κατάληψης των δορυφόρων και άλλα σχετικά. Καλά θα κάνουμε, εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε μια ικανότητα σε αυτά τα πράγματα, αλλά αν θέλουμε να παραμείνουμε μπροστά, θα πρέπει να κάνουμε τη σχετική προσπάθεια. Και η έκκλησή μου είναι, όχι μόνο για τον προπολογισμό του 2019, αλλά ιδίω στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να ενισχυθεί το πρόγραμμα COSME. Και θα παρακαλέσω τον πρόεδρό μας Μπούσεκ να κρατήσει την αρμοδιότητα εδώ στην Επιτροπή Ήτρε γιατί πρόκειται για έρευνα, πρόκειται για πολιτική βιομηχανία και ε, σε εμά ανήκουν οι αρμοδιότητε αυτέ και πρέπει να τι συνδιαμορφώσουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ, κύριε Σάρφ. Η κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Επίτροπε και εσείς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν έχω να κάνω σχόλια. Ευχαριστώ πολύ για την υποβολή των προγραμμάτων που αποτελούν μια εξαιρετική βάση επί της οποίας μπορούμε να διεξαγάγουμε σχετικές συζητήσεις. Οι δύο ερωτήσεις για το πρόγραμμα για το διάστημα και ιδίω για την δομή διαχείρισης. Είπατε ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός διαφορετικών οργανισμών, θεσμών που διαχειρίζονται τα διάφορα διαστημικά προγράμματα και ότι τελικώς είναι, υπάρχει κάποια σύγχυση. Η ΙΣΑ, η GSA, ο Frontex εν μέρη, ένσα, ενίσα και ούτω καθεξής. Είναι καλό λοιπόν, είναι καλή η πρότασή σας να είναι μια πιο διαρθρωμένη ε, δομή. Πώς όμως σκέπτεστε να το οργανώσετε. Μιλείτε και για ένα νέο οργανισμό για τα διαστημικά προγράμματα. Ο οργανισμός αυτός ε, θα συγκεντρώσει αρμοδιότητες και από άλλους λαμβάνοντας τις από άλλους και πώς θα διαμορφωθεί η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΖΕΣΑ και ΕΣΑ στο μέλλον Ευρωπαϊκής, ε, Ευρωπαϊκού ε, Οργανισμού Διαστήματος. Επιχειρησιακά πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Δώστε μας κάποιες ιδέες γιατί θα με βοηθήσετε έτσι και να μπορώ να κρίνω τις προτάσεις αυτές. Πάλι για το πρόγραμμα του διαστήματος, η χρήση των συνεργειών, synergies, για τον μη στρατιωτικό τομέα και τον τομέα της άμυνας. Ερώτηση. Πώς θα γίνει, πώς θα διαμορφωθεί, ποια πράγματα κινούνται ήδη. Και όπως είπαν οι συναδελφοί μου προηγουμένως, σε, σε σχέση με την χρηματοδότηση δηλαδή, νομίζω θα χρειαστούμε πολύ περισσότερα εκεί για τον τομέα αυτό. Πολύ περισσότερα κονδύλια δηλαδή που να ενταχθούν στο πολιτευστημο δημοσιονομικό πλαίσιο από ό,τι έχουμε κάνει τώρα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο Μπούσεκ. Δεν έχω άλλου που να ζητούν το λόγο. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν να συνεχίσω αυτό που είπε η κυρία Νίπλερ πριν από λίγα δευτερόλεπτα, από τη δική μου σκοπιά θεωρώ ότι θα είναι σημαντικό να μπορέσουμε να προωθήσουμε την, διαστημική, την ευρωπαϊκή διαστημική στρατηγική, να την κάνουμε γνωστή στη νέα γενεά, γιατί αν συγκρίνουμε την κατάστασή μας στην Ευρώπη με άλλες χώρες και με την Κίνα ακόμη, είναι, ότι καθίσταται πολύ σημαντική η πρόβαση αυτής της στρατηγικής, γιατί αφορά ολόκληρη τη βιομηχανία μας. Ένα θέμα είναι αυτό. Άλλο θέμα είναι για το νέο πρόγραμμα ενιαίας αγοράς για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμά μας COSME ήταν μια σταθερά των τελευταίων δέκα ετών. Οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις γνώριζαν καλά τι συμβαίνει. Τώρα όμως έρχεται μια νέα προσέγγιση. Θα θέλαμε κάποιες συμβουλές για τα πολλά εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεών μας. Τι να αναμένουν και να αναμένουμε. Πώς θα χρηματοδοτηθεί το σύνολο του προγράμματος. Ως τώρα τα πράγματα ήταν εύκολα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι γνωρίζετε ότι σε τέτοιες επιχειρήσεις συνεργάζονται 10, 15, 20, 50 άτομα. Να φτιάξουν κάτι το νέο, μια νέα πρόταση και μια νέα προσέγγιση στη χρηματοδότηση, ωστόσο αυτά είναι πολύ δύσκολα και περίπλοκα πράγματα. Τι να αναμένουμε λοιπόν, κυρία ε, Επίτροπε, σε ό,τι αφορά την νέα χρηματοδότηση. Αυτά είναι κρίσιμα πράγματα για πολλά εκατομμύρια, όπως είπα, Ε. Δεν βλέπω άλλου να ζητούν το λόγο, άλλου συναδέλφου. Παρακαλώ, κύριε Επίτροπε, να λάβει το μικρόφωνο και να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όλου σα ευχαριστώ για τι παρατηρήσει Γενικώ, ήταν με θετικό πνεύμα και καταλαβαίνω ότι προσπαθούν κάποια θέματα και εγώ τα είπα αρκετά γενικόλογα ε, βέβαια τα έχουμε ξανασυζητήσει για την πολιτική διαστήματος αλλά θα ήθελα να απαντήσω σε όλους και επίση όσο συντομότερα δυνατόν και όταν επίσης συζητήσουμε τον προπολογισμό να δούμε τα θέματα ε, ο καθένας χωριστά ή το κάθε θέμα χωριστά τέλο πάντων. Δύο-τρει εξ αυτών ρώτησαν για τον ε, ρυθμό που προχωρούμε, γιατί τόσο γρήγορα. Μα είναι γενικότερο το θέμα. Στην προηγούμενη θητεία η Επίτροποι ήθελαν από την 1η Ιανουαρίου να αρχίσει να ισχύει ο προπολογισμό, 1η πρώτου δηλαδή του 2021 προκειμένου. Οπότε για κάθε πρώτη τη Επιτροπή θέλουμε να υπάρχει το ίδιο διάγραμμα. Εξού και αυτό ο ρυθμό. Βεβαίω υπάρχει μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση, βεβαίω και αυτό ε, κατοχυρώνεται από την πρόταση. Παντώ το πιο σημαντικό είναι ότι εάν δεν έχουμε τέτοιο ρυθμό, τέτοιο χρονοδιάγραμμα, τότε χάνεται η ευκαιρία χρηματοδότησης από την αρχή του επομένου προϋπολογισμού. Ξέρω επομένω ότι πάμε κάπως βιαστικά. Δεν έχουμε πρακτική εμπειρία, αλλά βέβαια ε, έχουν γίνει διαπραγματεύσεις, συζητήσεις που έχουν βοηθήσει. Αλλά να γιατί προχωρούμε τόσο βιαστικά και είναι πιο σημαντικό να υπάρχει προϋποδότηση, να υπάρχει οργανισμός, όλα όσα χρειάζονται πριν την έναρξη του επομένου του δημοσιονομικού πλαισίου, οπότε να ε, χάσουμε την ευκαιρία χρηματοδότηση. Αλλά βέβαια η αξιολόγηση προβλέπεται και προχωρούμε από τη βάση των όσων γνωρίζουμε σήμερα. Επίσης, ταυτόχρονα συζητούμε τα προγράμματα. Τι ισχύει για αυτά και για το επόμενο πολιτές πλαίσιο και συζητούμε και τη σχέση με το EIDP που ήδη ισχύει, επί τη βάση των όσων υπόγονων τα κρατη και αυτά όλα βοηθούν. Αλλά βέβαια είναι κάτι όλος νέο ως πρόγραμμα και όλα τα δεσμικά όργανα και οι εταιρείε. Και τα κρατημέλη πρέπει να προσαρμοστούν και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όσον αφορά την συγχρηματοδότηση. Είπε 60% ο κ. Κρασνοντέμψικη να διευκρινίσουμε ότι θα υπάρξει πλήρες χρηματοδότηση 100% δηλαδή πριν τα πρωτότυπα για την φάση της έρευνας. 20% για το πρωτότυπο και άλλα 8 μετά. 80 συγγνώμη. 80-80% μετά. Γι' αυτό λέμε μήπως πάει 60. Πάντως αυτά προβλέπει πρόταση. 120 συν 80. Βεβαίω και αυτό είναι περιορισμένο γιατί είναι τα εξαπλάσια των όσων προβλέπει τώρα το πρόγραμμα και ε, το πλαίσιο η IDP για άμυνα δεν είναι πάρα πολλά, αλλά αυτό που θέλουμε να εξασφαλίσουμε να υπάρχει αποτελεσματικότητα καινοτομία, ε, εργασία Σε αυτά εστιαζόμαστε και ε, κράτη-μέλη αυτά τα θεωρούν θετικά και η βιομηχανία. Ακόμα και το 20% για τη φάση του πρωτοτύπου είναι καλοδεχούμενα. Δεν ξέρω τι θα βγει από τις διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα, αλλά έχουμε ακόμα 30 δις, οπότε τα 900, αυτό είναι διαφορά 900 εκατομμύρια. Τώρα ε, για τις χώρες μέλη του ΕΟΧ πρέπει να συμμορφωθούν με τους κανόνες της ενίας αγοράς. Συγκεκριμένα συζητώ το θέμα της οδηγίας ε, για τις ε, συμβάσεις και διαγωνισμούς. Υπάρχουν οι διατάξεις ασφαλείας και όλα αυτά κάνουν αυτές τις χώρες επιλέξιμες. Όμως θα πρέπει να συμμετέχουν στην χρηματοδότηση ακριβώς όπως ή αδίποτε χώρα μελός. Τώρα όσον αφορά τα έργα προγράμματα ΠΕΣΚΟ. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με την ε, Φεντρίκα Μοντερίνη και τον Επιτρόπο Μπούλτς των μεταφορών ούτω ώστε να υπάρχει κάποια λογική συνέπεια μεταξύ των επιμέρους προγραμμάτων. Γι' αυτό και είπαμε, γι' αυτό το 10% αύξηση της ε, συγχρηματοδότησης, εάν πρόκειται για κάποιο έργο, πρόγραμμα και πά. της μόνιμης διαθρωμένης συνεργασίας. Αυτά εφόσον κινούμεθα στο πλαίσιο επομένως της ΠΕΣΚΟ. Και αυτό πάει στην ερώτηση τη κυρία ε, Γκροστέτ για την κοινωνική προσέγγιση και γιατί να ισχύει η ειδική πλειοψηφία. Αυτό είναι ο σκοπό μου. Υπάρχει συνεργασία, αποτελεσματικότητα, να πιάνω το από περισσότερο επομένω τα χρήματα του δημόσιου κορδόνα στην Ευρώπη και πρόκειται για αποφασιστικό, αποφασιστική φάση όπου τα κράτη-μέλη αποφασίζουν για τι προτεραιότητε. Εκείνα αποφασίζουν ε, τι θα γίνει με το πρόγραμμα αύξηση των δυνατοτήτων μα, εδώ που κάνει η κυρία Μογκερίνη και κατόπιν θα κρυθεί το καθηγημένο πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσως προτρέχω τώρα, και κάποιε ερωτήσει θα απαντήσουμε μετά. Οπότε έχουμε αυτή την άμεση διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε θα κάνει αξιολόγηση η Επιτροπή για το πρόγραμμα, αλλά τα κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη αποφασίζουν. Δυνατότητες, προτεραιότητες, τα κράτη-μέλη. Τι άλλο έχουμε για να δω. Και έτσι θα εξασφαλίσουμε αυτή την κοινοτική προσέγγιση που αναφέρατε για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, EDA. Ε, θα έχουμε πολύ στενή συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Ο οργανισμός αυτός θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο, ανάντι, δηλαδή στα πλαίσια συνεργασίας με το, τα κράτη-μέλη για να οριστούν οι προτεραιότητες των ικανοτήτων, αλλά και κατάντι, ε, γιατί θα διαχειρίζεται συγκεκριμένα σχέδια. Τα κοινοτικά κονδύλια όμως, εξού και η άμεση διαχείριση, ε, η διαχείριση λοιπόν των κοινοτικών κονδυλίων θα γίνεται με βάση τους κοινοτικούς κανόνες και άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι φυσικά εγώ προσωπικά, ο διάδοχός μου, ο θα είναι αρμόδιος για τη διαχείριση των κοινοτικών κονδύλιων. Για την ενδιάμεση αξιολόγηση μίλησα ήδη. Για τις εξαιρέσεις. Πολύ σημαντικές ερωτήσεις για τις εξαιρέσεις. Ήταν και η πιο χρονοβόρα διαδικασία στον τριημερή διάλογο, η συζήτηση των εξαιρέσεων. Εγώ ήμουν ανέκαθεν της, της θέσης ότι πρόκειται για κοινοτικά κονδύλια και θα πρέπει να ευνοούν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Δεν είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα γιατί έχουν πολλούς δεσμούς με τρίτες χώρες, πολλές επιχειρήσεις. Και η ίδια η βιομηχανία έθεσε το ερώτημα πώς θα συνεργαστούμε ε, και πώς θα αξιοποιήσουμε τους δεσμούς που έχουμε με τρίτες χώρες. Και γι' αυτό ευχαριστώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί ήταν πολύ δύσκολη η διαπραγμάτευση. Χρειάστηκαν 9 ώρες για τη συζήτηση μόνο αυτού του σημείου. Γιατί ήταν το πιο δύσκολο στις ε, τριμερείς διαλόγους ε, για, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης για την Άμυνα. Έχουμε δύο εξαιρέσεις. για τι ε, εταιρείε που έχουν ευρωπαϊκή έδρα, αλλά δεν υπάγονται στον ε, έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τις άλλες εταιρείε που έχουν έδρα αλλά δεν έχουν υπόκειται σε πλήρη α, κοινοτικό έλεγχο και θα πρέπει να πληρούν τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, ασφάλεια εφοδιασμού. Δεύτερον, προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών ή των πληροφοριών των θωρακισμένων και όλα τα συναφή και ε, σεβασμός των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στην Ευρώπη. Αυτές είναι οι τρεις βασικές προϋποθέσεις ε, ε, και όλες οι κυβερνήσεις παγκοσμίω τέτοια μέτρα λαμβάνουν όταν ανοίγουν την αγορά άμυνα τους σε τρίτες χώρες. Αυτές είναι οι εξαιρέσεις που είναι ισορροπημένες και πολύ καλά οριοθετημένες. Έτσι επιτρέπεται η συνεργασία με τον ΝΑΤΟ χάρη σε εξαιρέσεις αυτές, γιατί μερικές χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ δεν είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καναδάς, Φερρυπίν. Την περασμένη εβδομάδα μάλιστα ήμουν ε, σε συνεδρίαση της ΝΑΚ και εκεί μας ε, εξήγησε το θέμα το ΝΑΤΟ. Παρόμοιες συνθήκε λοιπόν και προϋποθέσεις ισχύουν ε, και για τις ευρωπαϊκές χώρες όταν δραστηριοποιούνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπήρχαν κάποιες απορίες για τον οργανισμό. Η πρώτη είναι κάπως γενική και θα ήθελα να το πω καθαρά και εξάστερα. Δεν πρόκειται να ιδρύσουμε νέον οργανισμό. Το λέω στα ράτα. Έχουμε δύο ε, οργανισμούς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και το GSA, την Εποπτική αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS, του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης, που έχει έδρα στην Πράγα. Και θέλουμε απλώς να εξορθολογήσουμε τη διαχείριση, τη διακυβέρνηση των δύο ε, φορέων. Δεν έχουμε νέο οργανισμό, δεν έχουμε μεταφορά αρμοδιοτήτων. Πρόκειται για μια εξέλιξη γιατί όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα κατάσταση, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ περισσότερε αρμοδιότητε από ό,τι στο παρελθόν για τα προγράμματα του διαστήματο. Περί αυτού πρόκειται και τίποτα παραπάνω. Φυσικά, η κατάσταση για την εποπτική αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS είναι κάπω δύσκολη, ίσως ό,τι αφορά του μισθού και το λειτουργικό κόστο και η κατάσταση είναι κάπω δύσκολη. Δεν αυξάνουμε τον προπολογισμό ε, του οργανισμού, αλλά στα προγράμματά μας προτείνουμε να αυξηθεί το λειτουργικό κόστος για, τα, για να καλυφθούν τα νέα καθήκοντα, δηλαδή να αυξηθούν οι μισθοί, να καλυφθούν οι μισθοί και τα, το λειτουργικό κόστος ε, της εποπτικής αρχής που εδρεύει στη Πράγα, του GSA, της εποπτικής αρχής για το Ευρωπαϊκό GNS. Τώρα, πρόσβαση στο διάστημα. Και πάλι θα ήθελα να είμαι σαφής και δίκαιη γιατί αυτή ήταν η θέση που έλαβα από την αρχή της κοινοβουλευτικής, από την αρχή της θητείας μου, αυτόνομη πρόσβαση της Ευρώπης στο διάστημα. Και άρα χρειαζόμαστε γι' αυτό ευρωπαϊκούς εκτοξευτήρες και έχουμε και ένα ειδικό άρθρο στην πρόταση που καλύπτει αυτή την προτεραιότητα. Και προβλέπουμε δύο βήματα. Καταρχήν, συγκέντρωση της ευρωπαϊκής ζήτηση για τους εκτοξευτήρες που ανέφερε η κυρία Γκροστέτ και για την Αριανέξη και για το Vega C ε, και επίσης πιθανότητα να διαχωριστεί ένα κονδύλιο για την προσαρμογή των χερσαίων υποδομών. Αυτό προβλέπεται στην πρόταση, ειδικά και σαφώς. Κύριε Μαχτά, όπως σχεδόν πάντα συμφωνώ μαζί σας. Γιατί είμαι σαφής. Έχουμε ευρωπαϊκά κονδύλια, άρα θα πρέπει αυτά να ε, ωφελούν τις ευρωπαίες επιχειρήσεις και να μας επιτρέψουν να καλύψουμε τα τεχνολογικά κενά και να αυξήσουμε την καινοτομία αν χρησιμοποιήσουμε κοινοτικά κονδύλια για την ανάπτυξη τεχνολογίας, δεν θα πρέπει αυτή η τεχνολογία μετά να μεταφερθεί σε τρίτες χώρες. Και επίσης, αν δεν υπάρχει θεγράμμιση με του στόχου, να μπορούμε να ανακτούμε, να διεκδικούμε πίσω τα κονδύλια που επενδύσαμε, εφόσον δεν συνάδουν ε, ε, οι πορείε του με τους στόχου. Τώρα και ένα άλλο πιο προσωπικό σχόλιο. Αλλά επίτροπος είναι, δεν μπορεί να είναι και πολύ προσωπικό το σχόλιο. Ίσως ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και εσεί, στο μέλλον, το νέο κοινοβούλιο, θα πρέπει να ε, εξετάσουμε νέου κανόνε ανταγωνισμού, γιατί έχει σχέση με αυτό που συζητούμε τώρα. Και εκεί επίση συμφωνώ μαζί σα. Γιατί εμεί θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με τι δύο εξαιρέσει και με τι τρει προποθέσει για να διαφυλάξουμε την τεχνολογία να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ό,τι επιτύχουμε με τα ευρωπαϊκά κονδύλια να παραμείνει στην Ευρώπη αλλά γενικώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ξανασυζητηθούν οι κανόνες ανταγωνισμού στην Ευρώπη, γιατί δεν ευθυγραμμίζονται με τους κανόνες ανταγωνισμού που ισχύουν διεθνώ. Αλλά αυτό είναι περισσότερο προσωπικό σχόλιο, μια και είναι εκτός του χαρτοφυλακίου μου το θέμα του ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικέ δορυφορικέ επικοινωνίε, το πρόγραμμα GovSatcom εντάσσεται στο πρόγραμμά μας για το διάστημα. Εκεί προβλέπουμε πολύ μεγαλύτερη διασύνδεση με την άμυνα. Και έχουμε πλήρη ευελιξία εδώ. Θα έχουμε και νέες δημοσιονομικές γραμμές στο πρόγραμμα του διαστήματος για τα θέματα αυτά. Ε, μαζί με το κλίμα. Τι άλλο, τι άλλο και η ασφάλεια που είναι κάτι πολύ καινούριο στο πλαίσιο του διαστήματος. myself in those notes, but I think uh, governance, uh, I think I said. Για τη διακυβέρνηση. Συνεχίζουμε τις επικοδομητικές ε, συζητήσεις με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος που θα πρέπει και αυτός να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση και ο οργανισμός μας χρειάζεται και εμείς χρειαζόμαστε τον Οργανισμό Διαστήματος. Γιατί δεν έχουμε άλλο θεσμικό φορέα στην Ευρώπη με τόσο πλούσια πείρα, τεχνογνωσία και εμπειρία ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί σωστά τα κονδύλια μας και τα προγράμματά μας στο μέλλον. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν πρόκειται για επανάσταση, revolution, αλλά για εξέλιξη, evolution. Για το πρόγραμμα COSME, ίσως ε, έγινε μια παρεξήγηση. Ξέρω ότι το πρόγραμμα COSME θα μετανομαστεί, αλλά το περιεχόμενό του δεν θα αλλάξει. Το COSME θα παραμείνει με ένα δισεκατομμύριο ευρώ προϋπολογισμό. Στα πλαίσια των 4 δισεκατομμυρίων του προγράμματος για, ε, νέα αγορά, για το νέο πρόγραμμα για την νέα αγορά, το 1 δισεκατομμύριο θα πάει για το πρόγραμμα που λεγόταν COSME παλιά. Εγώ φταίω ίσως για την παρεξήγηση, γιατί το γνωρίζω από, το, ξέρω από την αρχή. Το πρόβλημα κόσμου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν συνδέεται με το γνωρίζοντα ή με πολύ συζητημένη έρευνα. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και έχει ε, αξιολογηθεί πολύ θετικά. Γι' αυτό δεσμεύτηκα ότι θα παραμείνει και αυτό θα γίνει. Δεν πρόκειται να εξαφανιστεί ή να ε, συγχωνευτεί με τίποτα άλλο. Το πρόγραμμα θα παραμείνει αμετάβλητο με εξαίρεση στο όνομά του. Τίποτα άλλο ή απάντησα σε όλα. Ευχαριστούμε. Άπειρα τα θέματα, αλλά και τα προγράμματα που πρέπει ένας επίτροπος να διαχειριστεί. Πολύ μεγάλη υπηρεσία σας και σας ευχαριστούμε για την συνεργασία. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, δεν θα αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε η κυρία Βιενκόφσκα. Α, μου είπαν ότι υπήρχε κάτι για την ιστορική γενετικότητα και για την διασύνδεση και τη συνεργασία. Ε, βέβαια, είναι πάγια η συνεργασία με τον Επιτρόπο και το πιο σημαντικό για τώρα και για την Επιτροπή και για τα κράτη-μέλη που έχουν κατεβάσει πολλές ιδέες είναι να υπάρχει ένα τέτοιο δίκτυο δρόμων που να είναι επιλέξιμο για την στρατιωτική κινητικότητα. Αυτό και θα προχωρήσουμε και σε άλλες ιδέες. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για τη δουλειά σας και για την προετοιμασία όλων αυτών των σημαντικών προγραμμάτων για την πραγματική οικονομία, για την αισθημική στρατηγική, για τη αισθημικά ε, προγράμματα. Είναι πραγματική οικονομία Ευχαριστούμε πολύ και πάλι Επίτροπε που ήρθατε. Εμείς θα συντάξουμε το σχέδιο έκθεση, στον Ιούλιο θα είμαστε έτοιμοι, όπως έχουμε υποσχεθεί. Και ως Ήτρε θα συνεργαστούμε στενά με την γενική σας διεύθυνση, αλλά η προσωπική επαφή μαζί σας είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι, ναι, και εγώ περιμένω πώς και πώς να τα ξαναπούμε. Σε 8 μήνες θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Ρωμανική Προεδρία. Αυστριακή και Ρωμανική Προεδρία. Uh, uh, dear friends, next point Α έρθουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξής μας που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον για μένα. Πρόκειται για εργαστήριο για την Βρετανική αποχώρηση και την πολιτική ICT. Ε, ελπίζω ότι έχετε λάβει το έγγραφο που σας δείχνω και θα αρχίσουμε σε λίγα λεπτά. Έχουμε έναν θαυμάσιο εκπρόσωπο των νησιών, όχι όμως των Βρετανικών νησιών από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά των νησιών γενικά. ο κύριος Σον Κέλλη. Αγαπητέ φίλε, σας παρακαλώ να προεδρεύσετε του πολύ σημαντικό αυτού εργαστηρίου. Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις του Brexit στις πολιτικές ICT. Δηλαδή για τις τεχνολογίες πληροφορικής και τεχνολογίας.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 Καλά λοιπόν κυρίες και κύριοι, με μεγάλη μου χαρά αντικαθιστώ τον ε, αξιοσέβαστο πρόεδρό μας Ζέρζι Μπούζεκ και έχω την χαρά να προεδρεύσω του σημαντικού αυτού εργαστηρίου Βρετανική αποχώρηση και πολιτικές για τις τεχνολογίες πληροφορικής και, τεχνο... και και ε, επικοινωνίας δεν μπορεί κανείς να αποφύγει. Το Brexit θα δούμε τώρα. Έχουμε πολύ ε, ικανούς ομιλητές που ε, θα σας ε, κάνουν σχετικές παρουσιάσεις και θα έχουμε και περίπου 10 λεπτά μάλλον θα από τα πρόσωπα αυτά και ως συνήθως θα έχουμε και την ευκαιρία τα μέλη μας να προβούν σε σχόλια ή σε υποβολή ερωτήσεων. Περίπου μια μισή ώρα έχουμε προβλέψει για αυτά. Θα δούμε πόση ώρα θα χρειαστούμε. Ο πρώτος λοιπόν για σήμερα το απόγευμα είναι ο Τζέι Σκοτ Μακρούς που θα μας δώσει μια επισκόπηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων του Brexit και ενδεχόμενου τρόπου να προχωρήσει η Ευρώπη των 27. Ο Σκοτ Μάρκους είναι Senior Fellow, fellow σε πανεπιστήμιο και ανεξάρτητος πάροχος συμβουλών για τις ηλεκτρονικές τεχνολογίες. Έχει γράψει πολλά papers και έχει γράψει και βιβλίο, άρα καλός είναι εδώ ο πρώτος μας ομιλητής. Σκοτ Μάρκος, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η παρατηρήσεις μου θα θέσουν το πλαίσιο και για τις άλλες ε, παρουσιάσεις οι οποίες θα προχωρήσουν σε περισσότερες λεπτομέρειες για την πολιτική για τις τεχνολογίες αυτές. Εγώ λοιπόν θα τα πω όλα αυτά για να δούμε τώρα εάν μπορούμε να δούμε τις διαφάνειες. Ας αρχίσουμε αμέσως λοιπόν. Η επίπτωση της αποχώρησης της, Βρετανίας, της Βρετανίας η αποχώρηση της Βρετανίας θα έχει σημαντική επίπτωση στο Ηνωμένο Βασίλειο ίσως λιγότερε επιπτώσει στην Ευρώπη των 27, αλλά οι επιπτώσει στην Ευρώπη των 27 είναι ο στόχο μας σήμερα. Αυτά θα οδηγήσουν σε μείωση των επαφών μεταξύ επιστημόνων και ερευνητών μεταξύ της Ευρώπης των 27 και αυτών που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και λιγότερη συνεργασία και διάδραση. Και ένα άλλο στοιχείο έχει σχέση με την απώλεια οικονομικών, οικονομιών κλίμακος. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο και θα τα δούμε καθώς θα περνούμε τις διαφάνειες. Ελπίζω ότι κάποιες με θα εμφανιστούν στην οθόνη και στις οθόνες σας. Καλά λοιπόν, η μορφή που θα λάβει η αποχώρηση θα παίξει ρόλο και στις, ε, στην φύση των επιπτώσεων, συζητήσεις Υπάρχουν πολλές πιθανότητες πάντως, πολλές δυνατότητες. Φαντάζομαι διαβάζει τις ίδιες εφημερίδες όπως και εγώ. Και μία δυνατότητα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο να αποφασίσει να αναστρέψει την αποχώρηση. Βέβαια είναι ασθενής η πιθανότητα αυτή, αλλά υπάρχει. Και το να ενταχθεί στον, ε, στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθερών Συναλλαγών, στον Ευρωπαϊκό μάλλον Οικονομικό Χώρο, ε, δεν ε, είναι επίσης πολύ πιθανό, αλλά υπάρχει πάση περιπτώσει μπορεί να υπάρξει και μια σχέση όπως αυτή με την Ελβετία ή να είναι περιορισμένη σε μια Συμφωνία Ελευθέρων Συναραγών. Ή και να φύγει χωρίς απολύτως καμία συμφωνία. Είναι διαφορετικές οι πιθανότητες αυτές. Α, Γιατί Οι, οι επιπτώσεις εάν ε, ε, μπει σε έναν ε, ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο θα είναι σχετικά μικρές. Τα άλλα σενάρια όμως οδηγούν σε κάποιες διαφοροποίησεις, κάποιες αποκλήσεις ό,τι αφορά ε, την, ε, τις ρυθμίσεις, τις κανονιστικές ρυθμίσεις και τις πολιτικές. Θα σας εξηγήσω με λίγα παραδείγματα. Το ένα είναι η περιαγωγή, το άλλο είναι η μεταφορά προσωπικών δεδομένων και τα δύο αυτά θα επηρεαστούν. Υπάρχουν και πολλά άλλα. Αυτά όμως είναι από τα πιο προφανή παραδείγματα. Ο χώρος που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία ή ευκαμψία έχει σχέση με την πολιτική της έρευνα Εκεί πολλή ε, συντονισμό γίνεται μέσω του προγράμματο Horizon 2020. Και το πρόγραμμα αυτό είναι ανοιχτό όχι μόνο σε χώρε μέλη τη Ένωση, είναι διαθέσιμο και στα μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, EEA, όπω η Νορβηγία για παράδειγμα. Όλοι αυτοί συμμετέχουν. Έχει ανοίξει και στην Ελβετία, η οποία έχει διμερεί συμφωνίε και βέβαια είναι και στην ΕΖΕΣ, Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθερών Συναλλαγών και ανοίγεται και σε χώρες όπως και το Ισραήλ ή άλλες αναπτυσσόμενες χώρες όπου το Ισραήλ δεν έχει καμία άλλη ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι όμως συνδεδεμένη χώρα, συνδεδεμένη χώρα ε, στο πρόγραμμα Horizon 2020 και χέρι των ίδιων προνομίων όπως και μια χώρα μέλος στις περιπτώσεις αυτές. Στα λίγα παραδείγματα που σας έδωσα, το ένα ήταν η περιαγωγή, το άλλο είναι η μεταφορά προσωπικών δεδομένων το, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρεί έως τώρα ότι για την περιαγωγή θα συνεχίσει με τις ίδιες ρυθμίσεις και μετά από την ε, αποχώρηση. Και οι operator λένε τα ίδια. Θα γίνει έτσι πράγματι δύσκολο να πει κανεί. Αυτό που μπορεί να ελέγξει το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι εσωτερικές, οι μεδαπές ρυθμίσεις. Δεν μπορούν να αποφασίσουν τις ε, χονδρικές πωλήσει μεταξύ, δεν μπορούν να βάλουν, μεταξύ δηλαδή χωρών, δεν μπορούν να βάλουν εκεί μια οροφή. Και το αντίθετο. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι οι πληρωμές αυτές μεταξύ χονδρεμπόρων εντό εισαγωγικών είναι κόστος. Και θα υπάρχει πρόβλημα εάν το κόστος αυτό υπερβαίνει τις τιμές. Υπάρχει ήδη πρόβλημα στην παιδαγωγή μέσα στις ε, χώρες της Ευρώπη των 27. Αν όμω ε, το κόστος μην γίνει μεγαλύτερο ανάμεσα σε αυτές και στην ε, Μεγάλη Βρετανία και βέβαια εταιρείε όπως η Vodafone μπορεί να απορροφήσει μεγάλο μέρος του κόστους αυτού. άλλε μικρότερες εταιρείε δεν μπορούν. Θα έχει λοιπόν το αποτέλεσμα αυτό οι network operators της Ευρώπης των 27 να έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική, δύναμη από αυτούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Και εγώ προβλέπω ότι λιγότερα προβλήματα θα σημειωθούν για τις ε, χώρες μέλη των 27 από ε, την περιοχή στο Ηνωμένο Βασίλειο παρά αντίθετα λόγω της μεγαλύτερης διαπραγματευτική ισχύω των operators στην ε, Ευρώπη των 27. Αν και όχι όλοι. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό να δούμε τώρα στις διαφάνειες μιας και φαίνονται. Το επόμενο θέμα που θέλω να καλύψω είναι οι μεταφορές προσωπικών δεδομένων. Τώρα υπό την ισχύ του νέου γενικού κανονισμού GDPR, προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταφέρονται με μεγάλη ελευθερία μεταξύ χωρών μελών και μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τρίτες χώρες βέβαια έχουν διαφορετικούς κανόνες και μπαίνουν ξεχωριστά στον GDPR. Γνωρίζουμε από το παρελθόν ότι οι διατάξεις ασφαλούς λιμένος που ε, χαίρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ανατράπηκε με απόφαση του δικαστηρίου του 2015, ε, το οποίο απέτησε να δημιουργηθεί κάτι που λέγεται privacy shield μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως τα γνωρίζουν πολλοί εκ των Ευρωβουλευτών, δεν έχει ακόμα αποδειχθεί αποτελεσματικότητα ε, του μηχανισμού αυτού. Αλλά πέραν αυτού, είναι ασφαλέ να πει κανεί ότι κάτι παρόμοιο μπορεί να αναμένεται και αυτή τη στιγμή αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εάν τεθεί το ίδιο θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οι παρόμοιε περιστάσει, οι παρακολουθήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πολύ διαφορετικέ από αυτέ τι Ηνωμένε Πολιτείε, θα δοθεί μάλλον μια παρόμοια λύση με αυτήν τη ε, ασπίδα τη προσωπική σφαίρα, privacy shield. Τώρα, η εμπειρογνωμοσύνη. Εκεί ο τρίτος ομιλητής μα, κ. Γιώβιτς, θα μιλήσει με περισσότερε λεπτομέρειε γι' αυτό. Το θέμα εδώ είναι ότι η regulatory expertise του Ηνωμένου Βασιλείου έχει παίξει σημαντικό ρόλο στι ρυθμίσει για, ε, το, για τις τηλεπικοινωνίες και θα λείπει τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να ενταχθεί σε άλλο βιασμό όπως RSPG. Είναι ε, δυνατόν να συνεχίσει να αναλαμβάνει το ρόλο αυτό ο οργανισμός Μπέρκ βάζοντας άλλες χώρες σε ρόλο παρατηρητού, όπως έχουν πράξει με την Ελβετία, που νομίζω ότι είναι λογικό, θα το παραδεχτούν όλοι. Μπορεί να διεξαχθεί λοιπόν διάλογος, ακόμη και αν οι ρυθμίσεις θα αποκλίνουν συν το χρόνο. Σε ό,τι αφορά περιορισμένη πρόσβαση για Βρετανούς ερευνητές και, και, και φορείς καινοτομίας, το θέμα εδώ είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σημαντική δύναμη προώθησης έρευνας και καινοτομίας και για θέματα, για παράδειγμα, ε, τεχνητής νοημοσύνης και εκεί η έλλειψή τους θα είναι αισθητή. Πολύ συντονισμός γίνεται μέσω του προγράμματος Horizon 2020. Εκεί υπάρχει προηγούμενο να συμμετέχουν άλλες χώρες ως συνδεδεμένα κράτη. Αυτό θα μπορούσε να συνεχιστεί και με το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε όλα τα σενάρια, εκτός ίσως από, το, από την πολύ σκληρή αποχώρηση που δεν είναι προς το συμφέρον ωστόσο ούτε ε, του Ηνωμένου Βασιλείου ούτε των χωρών μελών της Ένωσης. Ε, εν συνόψη η μορφή που θα λάβει το Brexit θα επηρεάσει όλες αυτές τις ρυθμίσεις. Εάν υπάρξει μια ρύθμιση ε, τύπου Νορβηγία δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Όλα τα άλλα σενάρια θα οδηγήσουν σε, αποσύνθεση, σε ρυθμιστική αποσύνθεση σε συγκεκριμένου τομεί. ο διάλογος και οι επαφέ μπορούν να συνεχιστούν για τις τεχνολογίες ε, επικοινωνιών. Αλλά αυτά θα φανούν μετά από το ε, Brexit. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε αρκετό, αρκετή τροφή για σκέψη και συζήτηση και τηρήσατε πραγματικά θαυμάσια τα όρια του χρόνου σας. Δεν θα είχατε κανένα πρόβλημα αν ήσασταν ευρωβουλευτής. Ας έρθουμε τώρα στον δεύτερο μιλητή, που είναι ο κύριος Μπάς Κότερινγκ, που θα αναπτύξει άλλες πτυχές της Βρετανικής αποχώρησης στην ψηφιακή καινοτομία αυτή τη φορά για ICT και TNO καινοτομία για τη ζωή. Είστε λοιπόν ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας ομιλήσετε. Ευχαριστώ. Ορίστε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ευκαιρία που μας δίνετε να πούμε λίγα λόγια για ένα αρκετά σημαντικό θέμα φυσικά. Μου ζητήθηκε να αναπτύξω τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου στα θέματα ψηφιακή καινοτομία και ποιε θα είναι οι συνέπειε του Brexit σε αυτή τη θέση. Περνάμε στην τρίτη διαφάνεια. Καταρχήν μια σύνοψη των σημείων που θα πραγματευτώ. Θα ξεκινήσω με μια επισκόπηση της θέσης του Ηνωμένου Βασιλείου στην ψηφιακή καινοτομία. Μετά ε, θα ασχοληθώ με το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων, τη έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη σε θέματα τεχνολογία, πληροφορία και επικοινωνία σε σχέση με αντίστοιχε προσπάθειε στην Ευρώπη. Και μετά θα μιλήσω για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τι διαδικτυακέ πλατφόρμε. Αυτά είναι τα τρία βασικά στοιχεία του πρώτου σημείου. Και μετά θα ε, κάνω μια επισκόπηση των βασικών συνεπειών τη αποχώρηση του Brexit από, αγορά, από την ενιαία αγορά και κάποια σημεία συζήτηση. Η επόμενη διαφάνεια τα λέει όλα. Παγκοσμίω το Λονδίνο είναι μετά το Silicon Valley και τη Νέα Υόρκη ε, ο τρίτος τεχνολογικός κόμβος και ε, είναι μακράν πιο αναπτυγμένος τεχνολογικός κόμβος στην Ευρώπη το Λονδίνο. Ε, ακολουθούν το Βερολίνο, το Άμστερνταμ και το Παρίσι, αλλά είναι πολύ πίσω. Σε ό,τι αφορά την ε, την πρόσβαση στη, στα χρηματοοικονομικά, την αγορά και τα ταλέντα, καθώς και την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, που με το Λονδίνο παγκοσμίω είναι ο τρίτος τεχνολογικός κόμβος. Οπότε, από αυτήν την άποψη, μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου έχουμε μια τέτοια ισχυρή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα πολύ ισχυρό ε, κλάδο fintech και δημιουργία. Και τέλο, και ίσω το πιο σημαντικό, είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια πύλη της Δυτικής Ευρώπης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και χάρη της αγγλικής γλώσσας, αλλά και της παρόμοιας κουλτούρας ε, των κοινών σημείων της κουλτούρας, της αντιμετώπισης του και των κεφαλαίων κινδύνου και της προσέγγισης που έχει σε θέματα τεχνολογικής καινοτομία. Η επόμενη διαφάνεια ίσως παρά είναι λεπτομεριακή, αλλά θα σταθώ σε λίγα μόνο σημεία. Πρόκειται για ένα μακροσκελή κατάλογο. Πρώτη στο κατάλογο είναι η Silicon Valley. Μετά έχουμε άλλους τεχνολογικούς και κόμβους καινοτομία στον κόσμο. Ε, βλέπετε αμέσω μετά τη Silicon Valley είναι η πόλη της Νέας και στην τρίτη θέση το Λονδίνο. Σε ό,τι αφορά την ε, πρόσβαση στη χρηματοδότηση για νεοφυείς επιχειρήσεις, για επεκτηνόμενες επιχειρήσεις. Είναι πραγματικά κόμβος καινοτομία στο Λονδίνο, στον κόσμο. Και η πρόσβαση στις αγορές στο Λονδίνο και στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικώ είναι από τους βασικούς παράγοντες που διευκολύνουν την κατάσταση. Το μόνο σημείο όπου κάποιες άλλες πόλεις στην Ευρώπη κάνουν, έχουν εξίσου πολύ καλές επιδόσεις είναι η πρόσβαση στα ταλέντα. Κάτι που δίνουν οι άλλε χώρε στο Λονδίνο και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ταλέντα. Υπάρχει μεγάλη ε, διακίνηση ταλέντων ε, και ατόμων και επιχειρήσεων και τροφοδότηση με ταλέντα της βρετανική αγορά. Φυσικά ε, η κατάσταση αυτή θα αλλάξει μετά τον Brexit, οπότε και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Άλλο σημείο που σχετίζεται και με τις παρατηρήσεις του Σκοτ Μάρκους για τις διάφορες μορφές που μπορεί να πάρει το Brexit. Ο, το Λονδίνο έχει και τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Δεν φαίνεται βέβαια αυτό από τον πίνακα. Αλλά σίγουρα το Λονδίνο έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, μαζί με τη Στοκχόλμη ίσως. Αλλά είναι σημαντικό ότι οι χώρες που είναι εκτός της Ευρωζώνης είναι αυτές που αναπτύσσονται με ταχύτερους ρυθμούς το Παρίσι έχει κάποια μικρή ανάπτυξη και το Βερολίνο αρκετά καλή. Αλλά το Λονδίνο έχει την πιο ισχυρή ανάπτυξη. Οπότε θα είναι και στο μέλλον ισχυρός παράγων ανάπτυξης. Άλλο θέμα. Ε, πάνε στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στις τεχνολογίες ε, και ε, στη και επειδή στη ρομποτική, στην υπολογιστική υψηλών ε, ε, επιδόσεων και μάλιστα και στην τεχνητή νοημοσύνη Έχουμε ηγετική θέση εκεί, πολύ καλές επιδόσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα μία βρετανική εταιρεία, η DeepMind, βρίσκεται πίσω από την επιτυχία της Google σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε έχει ε, έχει παρασκευάσει και chips και, ε, και ε, hardware, οπότε τέτοια εταιρεία θα είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Brexit. Και μάλιστα ήδη έχει εκτιμηθεί ως πάνω από 200 εκατομμύρια. Οπότε οι Βρετανικές εταιρείες είναι σε ηγετική θέση από αυτήν την άποψη της τεχνητή νοημοσύνης, υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και ρομποτική. Οπότε, χωρί πρόσβαση στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μείνει ακόμη πιο πίσω. Τώρα, οι μεγάλες πέντε επιχειρήσεις, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, ε, επενδύουν δαψιλό σε θέματα στρατηγικής, ε, σε ψηφιακά θέματα και σε ζητήματα αυτοπροσαρμοζόμενων μηχανών, machine learning. Και πολλές από τις εταιρείε αυτές, τις μεγάλες πέντε εταιρείε, τα πέντε μεγαθύρια, έχουν τα εργαστήριά τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και ε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι πιο κοντά έρχονται στην Ευρώπη αυτές οι μεγάλες πέντε εταιρείε. Μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου φτάνουν και στην Ευρώπη. και να σα δώσω κάποιε τάξει μεγέθου για, αυτές τις ε, για αυτά τα πέντε μεγαθύρια, ε, οι χώρες αυτές ετησίως έχουν περίπου 70 εκατομμύρια, όσο είναι ολόκληρος προϋπολογισμός, 70 δισεκατομμύρια πέρυσι μάλλον. Ε, ε, δηλαδή φτάνουν στον προϋπολογισμό του προγράμματος ορίζοντας. Και εδώ μιλάμε για τις εταιρείε αυτές κάθε χρόνο και τον προϋπολογισμό τους. Και μάλιστα αυξάνονται ραγδαία οι επενδύσεις των μεγάλων αυτών εταιριών. Οπότε είναι σημαντικό να μείνουμε κοντά στις δράσεις αυτών των ε, εταιριών του διαδικτύου. Ε, επίσης, ε, μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου και μέσω του ρόλου που παίζει έχουμε τις καλύτερες διασυνδέσεις με τις μεγάλες πέντε εταιρείε και τις μαζικές επενδύσεις που κάνουν σε θέματα διαδικτύου σε έρευνα στην ICT και σε ψηφιακή καινοτομία. Επίσης, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι προηγμένο ε, σε ό,τι αφορά τις ε, αγορές online. Ηγείται της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προηγείται ακόμη και των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα ποσοστού αγορών διαδικτυακών. Επίσης, η Άμα η Amazon επεκτείνει την παρουσία της στην Ευρώπη με ταχύτατους ρυθμούς και χρησιμοποιεί ως εφαλτήριο το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ε, το ασιατικό ε, ηλεκτρονικό εμπόριο έρχονται στην Ευρώπη μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα, για την, ενια... για την ψηφιακή ενιαία αν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, όταν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσει ίσω σημαντική πρόσβαση σε, στο ζωτικό οικοσύστημα των νεοφιών επιχειρήσεων, τις αγορές, την χρηματοδότηση, τα ταλέντα, γιατί εκεί είναι πολύ περισσότερες ε, οι νεοφυείς επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε αυτό το κλάδο των ICT. Επίσης, κάποιο τμήμα της καινοτομίας τους επηρεαστεί από νομοθεσίες όπως το GDPR, το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Το Ηνωμένο Βασίλειο ίσως ε, λειτουργεί πιο ελαστικά στον τομέα αυτό και μπορεί έτσι να ενισχύσει τη θέση του και γίνει ενδιαφέρον παράγοντας ε, και προσελκύσει πολύ περισσότερες εταιρείες και κυρίως ε, startups. Οπότε έχει με πιο ευέλικτη νομοθεσία μπορεί να ενισχύσει το Ηνωμένο Βασίλειο τη θέση του σε θέματα τεχνολογικών κόμβων. Επίσης, έχουμε μια νέα πρωτοβουλία για την τεχνητή νοημοσύνη που είναι κάπως ασαφής προς το παρόν. Υπάρχει κίνδυνο να μείνει πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σίγουρα θα χρειαστούμε πολύ σημαντική πρόθεση για να αντισταθμίσουμε ε, την απώλεια της πρόσβασης. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, είτε να αξιοποιήσουμε τους άλλους κόμβους που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θα πρέπει να κρατήσουμε υψηλό βαθμό έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, όπως είπε και ο Σκότ προηγουμένω. Θέλουμε ισχυρέ εταιρικέ σχέσει ε, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη με το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχει τόσο κεντρική θέση στον τομέα τη της καινοτομία, τη ψηφιακή καινοτομία. Αυτά ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Τόσα πολλά για να μπορέσουμε να προβληματιστούμε, να τα χωνέψουμε και στείλετε μηνύματα που δεν μας είχαν προβληματίσει προηγουμένω όσον αφορά τη θέση μας ως προς το νούμερο βασιλείο σε αυτόν τον τομέα. Προχωρούμε τώρα στον τρίτο ομιλητή, ο Ντόμαγκόι Γιούριεβιτς. Έτσι, έτσι ονομάζεστε, Ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος στο Συμβούλιο της ε, Ρυθμιστική Αρχή Κροατία για τι διαδικτυακέ βιομηχανίε και επίση έχει χρηματίσει αντιπρόεδρο του οργανισμού Μπέρεκ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σα. Στο χρόνο που μου αναλογεί θα σα πω για τι συνέπειε του Brexit για τις 27 χώρες μέλη. Νομοθεσία και ε, Σα Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία να έρθουμε εδώ και να μιλήσουμε. Στην ε, διαδρομή μου έχω εμπλακεί όσον αφορά την θέση της νομοθεσίας από πλευράς Μπέρεκος Ρυθμιστικής Αρχής και από πλευράς Κροατίας επίσης έχω ασχοληθεί με την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή. Οπότε για την παρουσίασή μου σήμερα θα προσπαθήσω να επισημάνω ποια θεσμικά όργανα, ποιοι οργανισμοί είναι σημαντικοί στον πράγμα την νομοθεσία και τη διαμόρφωση πολιτικής κατά τη γνώμη μου. Η Μπέρεκ είναι πολύ σημαντική αρχή όσον αφορά την εναρμόνιση της νομοθεσίας για όλη την Ένωση. Προετοιμασία της δουλειάς, επομένως, του Συμβουλίου και η κόκομ είναι πολύ σημαντική ως ε, ε, αρχή και έχουμε επίσης και φαρμοστικές ε, αρμοδιότητες, αριθμιστικές αν θέλετε. Οπότε λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν σε αυτούς τους οργανισμούς. Να δούμε όμως τι σημαίνει η σημερινή συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και τι δεν θα ισχύει όταν αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασιλείο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η εμπλοκή του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτούς τους τρεις τομείς. Αλλού έχει τη μορφή συνεργασίας μεταξύ ερτιμιστικών αρχών, διάδοση των αρίστων κανονιστικών πρακτικών σε κάποιους φορείς στη καθημερινή δουλειά, αλλού σε επίπεδο στρατηγικής, αλλά όπως βλέπετε εδώ είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το Ινωμένο Βασίλειο και άλλα κρατημέλη εμπλέκονται σημαντικά. Τώρα, ο τρόπος της εμπλοκής του Ινωμένου Βασιλείου ως κράτος μέλος. Να σας πω την προσωπική μου άποψη από την προσωπική μου εμπειρία. Στην ε, Μπέρεκ Επρόκειτο για την συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Τότε που προσχωρήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ σημαντικό γιατί χρειαζόμαστε την εμπειρογνωμοσύνη ε, όσον αφορά το καθημερινό μας ε, έργο. Επίσης υπήρχε το έργο που επιτελεί το σε επίπεδο ομάδων εργασίας όσον αφορά επίσης ε, τη σύνταξη εγγράφων και τον Βασιλό και άλλες χώρες ε, συμμετέχουν πολύ και τον Βασίλειο συνέβαλε στην ποιότητα των εγγράφων. Όσον αφορά τώρα το Συμβούλιο και την συνήθεια νομοπαρασκευαστική διαδικασία και σε αυτή την περίπτωση οι εκπρόσωποι των κρατών μελών εμπλέκονται. Είναι σημαντικό να υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά την αξιολόγηση της νομοθεσίας που θεσπίζεται και δημοσιοποιείται. Οπότε και οι συνομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διαθέτουν αυτήν την εμπειρογνωμοσύνη. Και από την αρχή, επομένω, τη προσχώρησή μα υπήρχε τέτοιο ρόλο για το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, όσον αφορά την Επιτροπή Επικοινωνιών, είχαμε εκτεταμένη συνεργασία, οι εκπρόσωποι των διάφορων κρατών μελών και δουλέψαμε, συνεργαστήκαμε για διάφορε προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτή την περίπτωση ήταν σημαντική πυρογνωμοσύνη για το καθημερινό μα έργο. Παρακάτω. Πάμε στι τρει διαφάνειε για να δούμε τι γίνεται με αυτά τα σενάρια στα ε, οποία αναφέρθηκε ο κύριος Σκότ Μάρκος. Αυτά τα τρία σενάρια είναι πρώτα πρώτα το σενάριο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ε, και το σενάριο σε σχέση με την ε, Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου. Τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να χαθεί, να λείψει από πλευράς αποχώρησης. Το πράσινο τσεκ σημαίνει ότι η κατάσταση θα μείνει όπως έχει τώρα το κόκκινο σημαδάκι σημαίνει ότι τα πράγματα δεν θα πάνε τόσο καλά. Οπότε όσον αφορά τη δουλειά μας, σχεδόν στο σενάριο ΕΟΧ, τα πράγματα θα μείνουν ως έχουν. ΕΟΧ, ε, ε, τους παρατηρητές, το, το Λίχτενστάιν, να λαμβάνουν μέρος σε εργασίες εκεί. και οι προτεραιότητε μπορεί ακόμα και αν δεν είναι. Μάλλον αυτοί που συμμετέχουν εκεί μπορεί ακόμα και αν δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προτεραιούν ομάδων εργασία. Τώρα στο Συμβούλιο. Πολλά θα αλλάξουν όταν πια δεν είναι κράτο μέλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα εμπλέκονται πια, δεν θα υπάρχει εμπλεγνωμοσύνη του. Ίσως συμμετέχουν σε κάποιες επιτροπές ως παρατηρητές, αλλά δεν θα συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων ως παρατηρητές, όπως είναι ο κανόνας, για τις διμερείς συμφωνίες. Τώρα ισχύει το ίδιο. Προναφέρθηκε και ο ρόλος της Ελβετίας που είναι παρατηρή στην Μπέρεκ, αλλά στην ε, Επιτροπή Επικοινωνίας και στο Συμβούλιο όχι. Τώρα στο σενάριο ε, Συμφωνίες ελευθερών μπορεί με τον Ρωμανό Βασίλειο. Όλα, όλα θα χαθούν. Δεν θα εμπλέκεται πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο πουθενά και για να κάνουμε μια σύνθεση στην τελευταία διαφάνεια βλέπουμε τώρα τι έχει αποφασιστεί, τι έχει αναγνωριστεί, θα είναι συνέπεια αλλά όλα εξαρτώνται από το τι είδους συμφωνία σύνδεσης θα επιλεγεί. Άρα, θα υπάρχει ε, συνέπεια επιρροή στη συνεργασία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών. Άλλωστε υπάρχει συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές ε, σε όλο τον κόσμο. Όσον αφορά τώρα την εμπλοκή της Δημιουργίας Αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Μπέρεκ θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες. Γιατί μια συμφωνία σύνθεσης υποβαθμίζει, αδυνατίζει τη συνεργασία. Τόσο όσον αφορά την ποιότητα της νομοθεσίας δεν θα έχουμε την ποιότητα από πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου γιατί δεν θα είναι πια κράτος μέλο. Όσον αφορά τώρα την Επιτροπή επικοινωνία τη ΚΟΚΟΜ δηλαδή, πάλι σε αυτό το σενάριο δεν θα έχουμε τη συμβολή της Βρετανίας και την ποιότητα. Επίσης, θα ε, υπάρξουν επιπτώσεις όσον αφορά τη διαδικασία εναρμόνισης των ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών για τη σχετική πολιτική όσον αφορά την περιαγωγή και όσον αφορά τον κανονισμό για την ε, ουδετερότητα και την ε, υλοποίηση της ψηφικής αγοράς. Γιατί αυτό είναι μια προσπάθεια τόσο ώστε να ωφεληθούν οι χρήστες. Έχουμε τη σχετική νομοθεσία σήμερα για την περιαγωγή. Κάποια πράγματα από αυτά που τώρα προβλέπονται θα αλλάξουν. Κατά τη γνώμη μου θα είναι συγκρίσιμη εκείνη η κατάσταση με την οικονομική κατάσταση των Ανατολικών Βαλκανίων. Γιατί υπάρχει συμφέρον να διευρυνθεί η σχέση του να συμπιεστούν οι τιμές, αλλά θα υπάρχουν θέματα νομικής βάσης. και σε οποιοδήποτε σενάριο. Αυτή θα είναι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και θα πρέπει κάθε φορά να προσέχει εάν θα υπάρχει παραβίαση των κανόνων του ΠΟΕ. Ό,τι κανονισμό και ενισχύει δεν θα είναι δεσμευτικό για το Ηνωμένο Βασίλειο. Για τελικού χρήστε και για τι εταιρείε του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, κατά την προσωπική μου γνώμη, η εμπειρογνωμοσύνη των εκπροσώπων του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν υψηλή ποιότητα και αυτό δεν θα υπάρχει πια. Αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί από τη συμβολή των άλλων κρατομέλων ή από άλλους οργανισμούς. Αυτό όμως δυστυχώς είναι εκτός θέματος όσον αφορά την παρουσίασή μου δυστυχώς. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιούριεβιτς. Περνάμε τώρα στην τελευταία παρουσίαση από τον κύριο Ζέραρ Παγκορέλ, που είναι καθηγητής οικονομικών επιστημών και θα, μιλήσει, θα μας μιλήσει για τις συνέπειες του Brexit ε, στην καινοτομία των υπόλοιπων 27 χωρών και την ανάπτυξη της ε, πέμπτης γενιάς 5G. Μάλιστα, ε, είχαμε και το περσινό έγγραφο για το ραδιοφάσμα. Έχετε το λόγο κύριε Πογκορέλ. Όπως γνωρίζετε, το 5G είναι μείγμα τεχνολογιών, προσφοράς υπηρεσιών και αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις βιομηχανίες όλου του κόσμου και βέβαια ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα από τα στοιχεία οικονομικής και βιομηχανικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επίπτωση της Βρετανικής αποχώρησης θα έχει μεγάλη σημασία. Θα έλεγα ότι παρόλο που είναι παγκόσμια τεχνολογία, έχουμε τα γεωγραφικά δεδομένα μεταξύ ε, Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης των 27 και αυτά τα γεωγραφικά δεδομένα μπορούν να ε, θεωρηθούν ότι δεν έχουν έπιπτωση, ίσως έχουν και θετική ή ίσως και αρνητική επίπτωση και εν πάση περιπτώσει κανείς δεν ξέρει, χρειάζεται περισσότερη μελέτη. αυτό το 5G, όπως είπα, είναι μείγμα. Έχουμε πρότυπα, έχουμε φορείς, δηλαδή εταιρείε που συμμετέχουν, έχουμε τη γεωγραφία, που βρίσκονται οι φορείς αυτοί που έχουν έδρα, που βρίσκονται τα βασικά κέντρα της γνώσης, της παραγωγής. Και τι σημαίνουν όλα αυτά για την συνολική οικονομία της Ευρώπης. Όσον αφορά τα πρότυπα, τα στάνταρτ, εδώ δεν προβλέπω αλλαγή, εκτός ίσως από την επιρροή κάποιων φορέων, κάποιων παικτών. Ε, 200 χώρες είναι παγκοσμίω, υπάρχουν και οι βιομηχανίες. Η 5G ως τεχνολογία ορίζεται σε διάφορα επίπεδα στο εθνικό, στο περιφερειακό. Στην Ευρώπη δεν είναι άμεσα η Ευρώπη, είναι η διάσκεψη των ευρωπαϊκών ε, εταιριών ή φορέων και είναι ο οργανισμός που έχει ε, θεσπίσει τα προηγμένα πρότυπα της 5G. Άρα δεν προβλέπω εδώ σημαντική επίπτωση εκτός βέβαια από την σχετική επιρροή των μεν και των δε, αλλά δεν αναμένω ε, σημαντικές επιπτώσεις. Όσον αφορά βέβαια την έρευνα και ανάπτυξη, εκεί η εικόνα είναι κάπως ε, διαφορετική. Εξέτασα τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν σχέση με το 5G με ε, στόχο τον Ρίτο το 2020 και είδα και ποιοι θα συμμετέχουν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα πανεπιστήμια, ε, σημαντική και πάρα πολλά, και σημαντικά και πολύ ε, ε, γνωστά πανεπιστήμια όπως το Σάρι, του Λονδίνου και άλλα έχουμε φορείς όπως το BBC, έχουμε operators της ε, κινητής τηλεφωνίας έχουμε και ερευνητικά κέντρα με βάση μέρα την ε, Μεγάλη Βρετανία γιατί εκεί πολλές πολυεθνικές εταιρείες και ιδίως για λόγους γλώσσας έχουν εγκαταστήσει τα ευρωπαϊκά τους ερευνητικά κέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και μεταξύ αυτών θα βρείτε και οι ιαπωνικές εταιρείες όπως η NEC, κορεατικές εταιρείες όπως η Samsung, ε, που ασχολούνται με τα ψηφιακά, ε, άλλες με αμερικανικές έδρες επιχειρήσεων αλλά ερευνητικά κέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν και ε, εταιρείε που έχουν μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα Βρετανικά πανεπιστήμια θα μείνουν. Βλέπουμε εμεί την Vodafone, η οποία είναι ο υπαριθμός, ένα ε, φορέας κινητής τηλεφωνίας και μεταφέρει το κέντρο βάρους των επιχειρήσεων της τώρα στην ε, υπηρετική ε, Ευρώπη και ο όμικρον 2 είναι ωστόσο μέρος του ομίλου τηλεφώνικα. Ποια θα είναι η στρατηγική της Τελεφώνικα, της Ισπανικής Τελεφώνικα, θα διαθέσει πόρους στη μονάδα της αυτή που είναι εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο ή θα τα μεταφέρει από εκεί. Και σε ό,τι αφορά τα οι soft centers στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ ενδιαφέρον. Τι θα κάνουν οι Ιαπωνικές, Κορεατικές, Αμερικανικές επιχειρήσεις θα παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή θα μετακινηθούν ως μπόνους για την Ευρώπη των 27 θα μεταφερθούν στις, θα μεταφέρουν δηλαδή τις εγκαταστάσεις τους και τις δραστηριότητε τους στην Ευρώπη των 27. Αυτά βεβαίως θα συζητηθούν από τη στιγμή που θα βγει το τζίνι από την μπουκάλα, από τη στιγμή που θα ανοίξει η πηξίδα της πανδόρας, θα δούμε ε, σημαντικές κινήσεις κατά πάσα πιθανότητα στον χώρο αυτό. Παρόλο που, όπως είπε ο συναδελφός μου προηγουμένως, μπορεί να ισχύσουν διαφορετικά καθεστώτα για τα βρετανικά ερευνητικά κέντρα ίσως ε, του τύπου του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σχέσεις με το Ισραήλ και ή με την Νορβηγία και το καθεξής. Αυτά όλα θα πρέπει να συζητηθούν και από τους διαπραγματευτές. Σε ό,τι αφορά τώρα τους βιομηχανικούς φορείς, το 5G έχει σημαντικές επιπτώσεις διάφορες βιομηχανίες, γιατί το 5G θα είναι η βάση για την ε, μεταλλαγή της κινητικότητας της ε, αυτοκινητοβιομηχανίας, πιθανότατα της ε, ε, βιομηχανίας παραγωγής ενέργειας και πιθανότητα και των υπηρεσιών υγείας. Θα δούμε, βλέπουμε μάλλον σε αυτή τη διαφάνεια εδώ τα λογότυπα των διαφόρων φορέων που είναι παγκόσμιας δραστηριοποίησης. Δεν είναι μοναχά ευρωπαϊκές, ούτε ειδικά ευρωπαϊκές. Η αυτοκινητοβιομηχανία, όταν καθιερώνει πρότυπα, αυτά υπερβαίνουν τα όρια μιας μεμονωμένης χώρας. Από την άλλη μεριά βέβαια σε ό,τι αφορά τις δημιουργούμενες υποδομές στην Ευρώπη θα είναι καλό εάν αυτοκινούμενα οχήματα ή οτιδήποτε άλλο να μπορέσουν να προχωρήσουν και πέρα από, το, από την ε, διόρυγα της μάχης, αλλά αυτά δεν είναι στα χέρια της βιομηχανίας. Θα δούμε τώρα και ποιοι είναι οι φορείς της λεγόμενης κάθετης βιομηχανίας. Είναι ενδιαφέρον διότι οι βιομηχανίες αυτές λειτουργούν και εφοδιαστικές αλυσίδες και ε, αλυσίδες δημιουργίας αξίας πέραν των συνόρων. Αυτό δεν έχει διαρευνηθεί πολύ. Μπορούμε να φανταστούμε ωστόσο ότι η παραγωγή μπορεί μέσα στα πλαίσια κάποιων σενάριων να επηρεαστεί σημαντικά. Και συχνά μιλούμε για το γεγονός ότι όταν βλέπουμε τα εργοστάσια του Νισάν στην νότια περιοχή του Λονδίνου για να φτιάξουν, στο Σάντερλαντ μάλλον, για να φτιαχτεί ένα αυτοκίνητο τα ανταλλακτικά τα θύματα του αυτοκινήτου δηλαδή, διαβαίνουν τα σύνορα μεταξύ Ευρώπη και Ηνωμένου Βασιλείου 27 φορέ. Η ανατάραξη αυτών των σχέσεων και η σημασία διατήρησης αυτών των αλυσίδων παραγωγής αξίας και εφοδιαστικής βεβαίως πρέπει να τεθούν υπόψη των διαπραγματευτών. Και σε ό,τι αφορά την διασυνδεσιμότητα. Αυτό εδώ έχει ενδιαφέρον. Αναμένουμε τη νέα αυτή γενιά τεχνολογίας 5G να βοηθήσει την μακρού αναμενόμενη ευρωπαϊκή πρωτοπορία στις ψηφιακές τεχνολογίες, γιατί το 5G θα καταστήσει ευκολότερη πιθανώς τη δημιουργία και νέων επιχειρήσεων για να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να θεμελιωθούν πάνω σε αυτό, να χτιστούν με τμήματα του διαδικτύου. Όσο περισσότερες λοιπόν οι γνώσεις, όσο περισσότερα δεδομένα μπορεί να συγκεντρώσει κανείς, τόσο το καλύτερο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έλεγα μάλιστα ότι όσο υψηλότερη η φραγμή μεταξύ Ευρώπης 27 και Ηνωμένου Βασιλείου, τόσο το χειρότερο και για τις δύο πλευρές και για όλους τους φορείς. Εάν τώρα δούμε ως συμπέρασμα τα θέματα. Ίσως να χάσουμε κάποια πράγματα από αυτό το όραμα του 5G, ότι δηλαδή μπορεί να παίξει ρόλο πρωτοπόρο η Ευρωπαϊκή Ένωση το 5G. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι άνθρωποι του οποίου συνομιλήσαμε έχουν σημαντικές επιφυλάξεις. Η κοινότητα της έρευνας και ανάπτυξης ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, βλέπουμε δηλαδή ότι οι συναδελφοί μας εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο λένε στις δημοσιεύσεις ότι οι ρυθμίσεις της Ένωσης θα μεταφερθούν, θα ενσωματωθούν στο Βρετανικό Δίκαιο, ό,τι και να γίνει. Άρα, μένει να παιχτεί ένα σημαντικό παιχνίδι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι διαπραγματευτές μας γνωρίζουν και οφείλουν να γνωρίζουν τις ενδεχόμενες επιπτώσεις. Σας ευχαριστώ. Sorry. Thank you very much indeed. again... Σας ευχαριστούμε θερμά και σε ευχαριστώ που τηρήσετε και το χρόνο σας. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις ε, για τις ε, πιθανές συνέπειες του Brexit στις τεχνολογίες ε, πληροφορίας, στην πολιτική για τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην Ευρώπη. Υπάρχουν σχόλια? Αν όχι, να αναφερθώ σε κάποια σχόλια ε, από τη σκοπιά της Ιρλανδίας που θα επηρεάσει ιδιαίτερα από τον Brexit. Αναφέρονται για τις σχέσεις ε, Ένωσης ε, και Brexit το ότι όλοι θα βγουν χαμένοι. Ποιος όμως θα βγει περισσότερο χαμένος αν δεν υπάρξει κάποιος συντονισμός, κάποια κατάλληλη συμφωνία για συνέχιση όσο γίνεται πιο όμοιας κατάσταση με τη σημερινή. Επίσης, όσον αφορά την περιαγωγή και τις σχετικές χρεώσεις που ισχύουν και αυτά που κατάφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποιος είναι πιο χαμένος στην περίπτωση αποχώρησης εάν δηλαδή δεν ακολουθήσουν τις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Επίσης, κάποια άλλα σημεία μου φάνηκαν ενδιαφέροντα και τις διάφορες συμφωνίες με Νορβηγία, Καναδά και άλλες. Αυτά πώς σχετίζονται με τον ορίζοντα 2020 αυτοδικίως. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει το νούμερο στο ορίζον 2020. Ε, μια που το Ισραήλ δεν είναι κράτος μέλος, αλλά καλύπτεται. Επίσης, κάτι το οποίο αναδεικνύεται ως θέμα συζήτηση είναι αυτό το οποίο αναφέρει ο κύριος Μπαρνιέ. Την επιλεκτική εφαρμογή, επιλεκτική ισχύει. με μονομένο θεμάτων. Από πολιτική πλευρά, αυτό το cherry picking, όπω λέγεται, για την Ένωση ή για τον Ομίλιο Βασίλειο, θα μπορούσε να είναι ιδεώδε. Αλλά αυτό πώ συντεριάζει με την προσπάθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει το ίδιο καθεστώ και με το να εξηγούν τα ίδια προνόμια. Επίσης, αυτό το πρίβαση shield που αντικατέστησε την αρχή του ασφαλούς λιμένος. Θα ισχύει για το νούμερο βασίλειο. Τι άλλο μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Α, λέμε το νούμερο βασίλειο είναι η πύλη προς τις ΥΠΑΑ. Το ερώτημα είναι, μπορεί να αντικατασταθεί αυτή η πύλη, γιατί το Εμενό Βασίλειο και το Λονδίνο συγκεκριμένα, πώς μπορεί να συνεχίσει να είναι πύλη προς τις είπα για την Ένωση, όταν δεν ανήκει σε αυτήν, ήταν μια αντίφαση. Ε, τώρα είπαμε, χθες το Λονδίνο έχει πάρει στο Στοχόλμη, το Βερολίνο και άλλες πόλεις. Οπότε θα υπάρξει προσπάθεια αυτών σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Οπότε θα συνεχίσει να πρωταγωνιστείς για τεχνητή νοημοσύνη το Ηνωμένο Βασίλειο. ισχυρή χώρα. Πρωταγωνίστρια σε αυτό τον τομέα με τις εταιρείε της. Τι θα γίνει, θα υπάρξει ψηρήγνωση αυτού του πρωταγωνιστικού ρόλου λόγω του Brexit. Αυτά, αυτά ήθελα να σας αναφέρω. Α, έχω και μερικά άλλα. Νομίζω ο κύριος Πόγκορα λέει ότι θα χαθούν τα πάντα σε επίπεδο οικονομίας. Και εσείς κάτι είπατε κύριε Γιώργιεβιτς. Αναφέρθηκαν οι εταιρείε στο Ηνωμένο Βασίλειο που μετά το Brexit θα μείνουν εκεί. Θα αλλάξει κάτι. η Μάλτα. Τι θα γίνει με τις εταιρείες. Είναι πολύ καλό το ότι έχουμε εδώ πέρα τις σημειώσεις από αυτά που είπατε και όταν τα μελετήσουν βουλευτέ θα ε, προκύψουν πολύ περισσότερα ερωτήματα. Οπότε τώρα εσείς έχετε τη σκητάλη για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. In direction. <clears throat> okay, uh, as far as the lose, lose... Σε ό,τι αφορά το ποιο βγαίνει περισσότερο χαμένο, μια και όλοι θα είναι χαμένοι. Νομίζω ότι πιο χαμένο θα βγει το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλοι θα βγουν χαμένοι, αλλά περισσότερο το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, τι κλάσμα του Βρετανικού εμπορίου θα πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστροφο, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και γι' αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο θα βγει περισσότερο χαμένο. Σε συγκεκριμένου τομεί θα είναι πολύ σημαντικέ και σοβαρέ συνέπειε. Και ένα κλάσμα του ΑΕΠ, του Βρετανικού ΑΕΠ, προέρχεται από τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Και ο κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί ναι, δεν υπάρχει αυτή η γέφυρα με τι Ηνωμένε ε, Πολιτείε, αλλά γιατί έχει και πολλά φορολογικά πλονεκτήματα και παραμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε σίγουρα πολλέ χρηματοπιστωτικές επιχειρήσει θα φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο με το, με Brexit και θα επηρεάσει σίγουρα τον κλάδο μια τέτοια διαφορά, γιατί πολλά Ινστιτούτα που βρίσκονται στο Λονδίνο έχουν θηγατρικές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είτε στην Ιρλανδία, το Άμστερνταμ μπορεί να βγει πολύ ωφελημένο. Και εκεί θα βγει χαμένο το Ηνωμένο Βασίλειο στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που είναι πολύ σημαντικός κλάδος της Βρετανικής οικονομίας. Σε ό,τι αφορά τα τέλη περιαγωγής και εκεί θα βγει πιο χαμένο το Ηνωμένο Βασίλειο. Και ένας από τους βασικούς λόγου είναι και πάλι ο αριθμό των Βρετανών πελατών που ταξιδεύουν στην ε, Ισπανία, στην Ελλάδα και ακριβώς η διαπραγματευτική θέση ε, των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι καλύτερη και η πιθανότητα να κρατήσουν τις ρυθμίσεις του, της περιαγωγής ακόμη και αν δεν τις διασφαλίσει πλήρως το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μεγαλύτερες. Πάντως ε, το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί και ότι επιθυμεί να διαφυλάξει αυτέ τι ρυθμίσει για την περιαγωγή. Αλλά πιστεύω ότι μάλλον το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει περισσότερα να χάσει από το Brexit. Σε ό,τι αφορά τη διαφορά του μοντέλου Νορβηγία ή Καναδά, τι είδου εμπορικέ σχέσει. Έχετε δίκιο, δεν θα πρέπει να είναι αυτόματη η συμμετοχή στον ορίζοντα 2020. Ε, υπάρχουν όμως διαφορετικές αποχρώσεις ως μέλος του ΕΟΧ και μέσω του κανονισμού του ΕΟΧ ε, μπορεί να συμμετέχει στο ορίζοντα 2020. Σε άλλες περιπτώσεις, ε, αν δεν υπάρξει καμία συμφωνία απολύτως ή αν συναυθεί μόνο συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, τότε θα επαφείται απολύτως στη διακριτική ευχέρεια. Και μηχανισμός είναι ότι συνάπτει ε, συμφωνία σύνδεσης όπου ε, συμβάλλει οικονομικά ανάλογα με τον ε, συντελεστή του ΑΕΠ ως προς το κοινοτικό ΑΕΠ. Και εκεί θα πρέπει να ληφθεί απόψη γιατί με πολλές χώρες που θα μπορούσαμε να έχουμε σχέσεις τώρα θα οι σχέσεις αυτές είναι περισσότερο ανταγωνιστικές ή περισσότερο συνεργασίας θα προτιμούσα και σε πολλά, με βάση πολλά σενάρια, θα, μάλλον θα ήταν συνεργα, συνεργασίες περισσότερο. Τώρα, ένα σενάριο που συζητήθηκε ελάχιστα είναι μήπως το Ηνωμένο Βασίλειο γίνει ένας ε, ανταγωνιστής low cost σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τέτοια περίπτωση σίγουρα το ορίζοντα 2020 δεν θα είναι αυτόματη επιλογή. Ε, πάντως ε, απεύχομαι την υλοποίηση αυτού του σενάριου. Σε ό,τι αφορά την ασπίδα ιδιωτικότητα, αν σκεφτεί κανεί το αριθμό των πολυεθνικών και των ομίλων που έχουν γραφεία και παραρτήματα και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ σημαντική η διασυνοριακή συνεργασία και μπορεί να έχουμε κάτι παρόμοιο με αυτό που ισχύει για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων. Θα έχουμε απώλειες που θα επηρεάσουν τη, τον ψηφιακό τομέα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των 27 και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και σίγουρα οι 27, με βάση όλα τα σενάρια, προτιμούν να, να καταλήξουν λύσεις που θα μοιάζουν όσο γίνεται το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Πάντως, μία δικαστική υπόθεση θα μάλλον θα έλεγε ότι χρειάζεται κάτι παρόμοιο με την ασπίδα της ιδιωτικότητας και ίσως καταλήξουμε σε πιο αυστηρές, αυστηρές διατάξεις από την ασπίδα ιδιωτικότητας που είναι σχετικά χαλαρή. Ε, θα χρειαστούν τις ρυθμίσεις που θα εφαρμόζονται καλόπιστα και από τις δύο πλευρές. Ε, πάντως, ε, ακόμη είναι ασαφής η θέση και της Αμερικανικής κυβέρνησης ως προς αυτό. Ποιο θα μπορούσε να αντικαταστήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στο ρόλο της πύλης ε, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, όπως είπατε και η Ιρλανδία και η Μάλτα είναι αγγλόφωνε χώρες ε, και φαντάζομαι θα είναι πολλές πια οι πύλες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί υπάρχουν πολλοί αγγλόφωνοι και στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία σίγουρα και έχουν και πολύ καλύτερα αγγλικά από τα δικά μου. Αυτά και δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι θέλουν να απαντήσουν επίσης. Θα ξεκινήσω με το ότι θα μπορούσε και τα, να χαθούν τα πάντα. εγώ εξέτασα τις συνέπειες στην Ευρώπη των 27 και την ε, συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, από τη σκοπιά της εμπειρογνωμοσύνης, και της κανονιστικής εμπειρίας. Πάντως, οι ζημίες θα είναι και από τις δύο πλευρές. Και όταν ένα ζευγάρι χωρίζει, χάνεται η επαφή μεταξύ των δύο συζύγων, πρώην συζύγων. Οπότε ε, δεν έχουμε την καθημερινή βοήθεια, τις καθημερινές γνώσεις και συμβουλές και φυσικά αν δεν υπάρχει συνεργασία, ποιο το νόημα να παραμείνουν οι δύο σύντροφοι μαζί. Δεν ξέρω ποια πλευρά θα υποφέρει περισσότερο πάντως από το διαζύγιο αυτό, από την αποχώρηση αυτή. Ε, νομίζω ότι αυτοί που θα βγουν περισσότερο χαμένοι είναι οι τελικοί χρήστες και από τις δύο πλευρές, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 και από το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί πριν τον κανονισμό ε, για την περιαγωγή ε, ε, του 2007 όλα ακολουθούσαν τις αρχές της αγοράς. Οπότε, επειδή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών όλα είναι θέμα κλίμακος, ίσως καταλήξουμε ρυθμίσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με κάποιες με, να είναι διαφορετικές με μεγάλες χώρες όπου υπάρχει ισορροπία μετακινήσεων είναι διαφορετικές από ρυθμίσεις με μικρότερες χώρες που είναι λιγότερες συναλλαγές. Και εκεί θα εξαρτηθεί ποιος βγαίνει α, χαμένος περισσότερο. Στην πατρίδα μου, έχουμε, στην Κροατία, έχουμε περισσότερους Βρετανούς τουρίστες. Οπότε αν δεν ισχύσουν πια κάποιες δεσμευτικές ρυθμίσεις, ίσως οι Βρετανοί τουρίστες που έρχονται στην Κροατία δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες όπως το κάνουν στην πατρίδα τους, αν δεν ισχύσουν τα τέλη περιεγωγής. Ε, πιστεύω λοιπόν σε τελική ανάλυση ότι οι καταναλωτές είναι αυτοί που θα πληγούν περισσότερο από τον Brexit. Και πάλι όμως θα είναι θέμα αριθμών και σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών ανάλογα με το εμπόριο που έχουμε μεταξύ του τον τουρισμό και το καθεξής. Ε, εκείνες θα συμφωνήσουν αν συμφέρει να κρατήσουν τις τιμές ε, στα τωρινά πλαίσια ή να τις αυξήσουν. Μάρκος, όπως θα είναι το ημεροδοσίλιο είναι τώρα η Ελέδια συμμετέχει στην Μπέρεκ, συμμετέχει στις στατιστικές της Μπέρεκ για την περιεγωγή, αλλά δεν συμμετέχει στο σύστημα και τελικά για την περιοχή περισσότερα οι καταναλωτές στην Ελβετία παρά οι Άγγλοι. Οπότε το θέμα είναι αν θέλει το φύγει αυτό η Αγγλία, το Ιωμένο Βασίλειο δηλαδή, αν θα τα καταφέρει. Κότερινγκ. Για το θέμα της πύλης προς τη είπα. Ε, ναι, αν γίνει το hard Brexit θα είναι δύσκολο να υπάρξει η, η πύλη δεν ναι, βέβαια δίνεται αγώνας να μην αποκλειστεί η ενία αγορά. Ε, αν, τα, χάσουν αυτό το οποίο έχουν σήμερα θα είναι ανόητο. Αν έχουμε soft Brexit, τότε θα μείνουν τα πράγματα ως ε, έχουν. Οπότε για τις ε, ξέχουσες ε, νεοφύης θα είναι πολύ σημαντικό αν μπορούν να κατασταθούν εκεί. Γιατί οι Άγγλοι έχουν τα λεφτά και το ταλέντο το έχει η Ευρώπη. Άρα θα είναι καταδικασμένοι η Βρετανία. Και για το 5G είναι πολύ σημαντικό το χρονοδιάγραμμα. Ε, εντάξει, θα χάσουμε τον ρυθμό εξέλιξης αν δεν συμμετέχει η Αγγλία, αλλά θα βρεθεί, θα βρεθεί κάποια λύση. Δεν μπορεί παρά να γίνει αυτό, θα ήταν ανόητο. Όχι, όχι, δεν είναι καλό για μας αν δεν γίνει κάτι τέτοιο. Και για την τεχνητή νοημοσύνη. Το ίδιο ισχύει. Το εύκολο είναι έρευνα ανάπτυξη. Οπότε θα υπάρχει στενή συνεργασία και δεν υπάρχει άλλο σενάριο για μένα. Θα συνεχίσει να υπάρχει στενή συνεργασία. Κύριε Πόγκρελ, για να κλείσουμε. Τελευταίος εσείς. Για το 5G. Την τεχνολογία. Η κλίμακα, η κλίμακα είναι το ζουμί. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι. Ακόμα και από το 12% του πληθυσμού ή τέλο πάντων να το δούμε πιο απλά το κομμάτι της αγοράς. Δεν είναι καλό αυτό για τους 27, ε, αλλά είναι ακόμα χειρότερο για το ημέρο Βασίλειο. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση η κλίμακα. Κατόπιν είναι το θέμα του γεωγραφικού παράγοντα. Νομίζω ότι ο γραφικό εξηγεί γιατί τόσοι φεύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο και πάνε στους 27. Δεν είναι καν θέμα χαμηλού παραγωγής. Δεν μπορεί να μείνει ηγέτης στο 5G, σε διάφορες συσκευές αντίστοιχες. Πού να ανταγωνιστούν οι Βρετανικές εταιρείε της Samsung και την Apple. Φεύγουν, φεύγουν οι έχονται τη γνώση την εμπειρογνωμοσύνη από τον Ηνωμένο Βασίλειο. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει και με το πιο πιθανό σενάριο. Και στις διαπραγματεύσεις που σίγουρα έχουν ένα παγκόσμιο βεληνικές να δούμε αν θα επιτρέψουμε αυτή την επιλεκτική συμπεριφορά όσον αφορά την ε, έρευνα. Και αν θέλουμε να συνεχιστεί η συνεργασία με τους ε, Βρετανούς συναδέλφους. Θα ήταν ένα δωράκι προς την κυβέρνηση της Βρετανίας που δεν θέλει να το κάνει η Ευρώπη. Άρα τελικά κατά πολύ εξαρτάται από το πόσο ε, ευφύης θα είναι οι διαπραγματευτές, τι παζάρι θα γίνει. Να, ε, είναι παράδειγμα του δίληματος που αντιμετωπίζουμε. Το Γαλιλαίο, το, ο στο πρόγραμμα. Το σύστημα Γαλιλαίος θα αποτελέσει αντικείμενο πολύ σκληρών αποφάσεων. Δύσκολο. Δεν κάποια δισεκατομμύρια η Βρετανία, αλλά παίρνουν 14 δις και λένε πόπο θα χαθούν όλα αυτά τα λεφτά για τους 27 αλλά βέβαια όσο πιο μεγάλο είναι ένα σύστημα δορυφορικό, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι. Και αν χάσουμε τον Γαλιλαίο ίσως, οι λόγοι να είναι πολιτική, είναι και θέμα άμυνας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ δύσκολε αποφάσεις. Διλήμματα, ανταλλάγματα, παζάρι. Κέλλη. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο Σον Κέλλη. Ευχαριστώ και όλου του εμπειρογνώμονε για τις τοποθετήσεις τους, πραγματικά πολύτιμες για τις συζητήσεις μας, μας δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθεί η συζήτηση. Και αποτελούν την βάση για τις συζητήσεις που θα διεξαγάγουν οι συναδέλφοι μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Μάρκους, κύριε Κόσεμικ, κύριε Γιούρεβιτς και εσείς κύριε Πόρεβελ, χαιρόμεθα πολύ που σας είδαμε σήμερα. Πράγματι καταβάλλατε σημαντική προσπάθεια. Νομίζω τα είπατε με τρόπο που όλοι μπορούν να καταλάβουν. Καλά, τα καταφέρατε. Αυτό δείχνει ότι είστε επιδέξει στις επικοινωνίες. Ερχόμαστε στο τελευταίο θέμα της ημερησία διατάξεως. Δεν υπάρχει άλλο. Η επόμενη συνάντηση στις 19 Ιουλίου 3 έως 6.30 και την επόμενη μέρα από το πρωί στις 9 έως 12.30 και 14 και 30 18 και 30. Εδώ διακόπτω τη συνεδρίαση και σας ευχαριστώ πολύ.